Σας παρακαλώ θα αρχίσουμε. Αρχίζει η συνεδρίαση της Επιτροπής. Έχουμε ένα σημαντικό απόγευμα μπροστά μας και θα προχωρήσουμε με κάποια ταχύτητα. Πρώτα έγκριση της ημερησίας διατάξεως και σας ε, πληροφορώ ότι στην συνάντηση των συντονιστών συζητήθηκε η κατάσταση κρίσεως που αντιμετωπίζουν πολλοί τομείς στην ε, Ευρώπη με τις πολύ χαμηλές τιμές, με τις δυσκολίες που προκύπτουν για όλους τους γεωργούς και όχι μόνο τους κτηνοτρόφους και γαλακτοπαραγωγούς. Αποφασίσαμε λοιπόν να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε δήλωση θα γίνει δεκτό το έτοιμά μας και θα διεξαχθεί συζήτηση για την διαχείριση της κρίσεως στην επόμενη ε, περίοδο συνόδου του ε, Στρασβούργου, 14 έως 17 Δεκεμβρίου. Εάν είστε σύμφωνοι, ε, εγκρίνουμε και τα πρακτικά, ενώ της 19ης Οκτωβρίου και της 10ης Νοεμβρίου. Θεωρώ ότι εγκρίνονται λοιπόν. Η σημερινή συνεδρίαση διοχετεύεται ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο. Η ακρόαση θα γίνει στην εβδομάδα της 11ης Ιανουαρίου 2010. Η επιβεβαίωση θα γίνει, προβλέπεται από την ε, ε, Ολομέλεια, στην εβδομάδα της 25ης Ιανουαρίου. Μετά από την σημερινή συνεδρίαση η οργάνωση των ε, παραγωγών βιολογικών προϊόντων, η ΦΟΑΜ, προσκαλεί σε διεξίωση μετά από την συνεδρίαση. Το δεύτερο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την οργανική αντιμετώπιση των τροφίμων την εποχή των κλιματολογικών αλλαγών. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα έχουμε πρώτη του μηνός και τίθεται πλέον σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό σημαίνει βαθύτατες αλλαγές για, την Ευρωπαϊκή, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την, και την Επιτροπή μας. Από σήμερα θα συναποφασίζει το Κοινοβούλιο για θέματα γεωργίας. Αυτό μας δίνει περισσότερες αρμοδιότητες Ταυτόχρονα βέβαια μας δίνει και περισσότερες ευθύνες. Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες αυτές και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε όχι μόνο για τον γεωργικό τομέα αλλά για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι ζητούν μια λογική κοινή αγροτική πολιτική που να διασφαλίζει τα τρόφιμα, την ανάπτυξη της υπαίθρου και φυσικά την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων αγροτών. Από σήμερα λοιπόν ξεκινά μια νέα διαδικασία και εύχομαι κάθε καλύτερο σε όλους. Στο σημείο 5. Πολιτική ποιότητα στα γεωργικά προϊόντα. Ο Τζακάβλος Κοτά εισηγητής. Σήμερα θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. Είναι πολλές οι τροπολογίες αυτές. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σκοτά και όλους τους κοιόδης εισηγητές που συνεργάστηκαν η έκθεση πρωτοβουλία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά με την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων έχει προκαλέσει έντονα προσοχή. Έχουν κατατεθεί πάρα πολλέ τροπολογίε και το αποδεικνύουν αυτό. Θα πρέπει να συζητήσουμε αμέσως λοιπόν το θέμα και ζητώ από τον Τζακάρλο Σκοτά να μας δώσει τις δικές του απόψεις για, το, για την κατεύθυνση την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Έχει το λόγο η συγητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι μια καλή ευκαιρία για να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους και το ενδιαφέρον που έδειξαν για τη συγκεκριμένη έκθεση. Εξέτασα όλες τις τροπολογίες οι οποίες κατετέθησαν και θα ήθελα να σταθώ σε κάποιες από αυτές. Considero favorevolmente l'emendamento numero 14 presentato dall'onorevole Lefort. Είμαι υπέρ της 11. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερασπιστεί τα ποιοτικά προϊόντα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ. Θεωρώ επίσης ότι είναι θετική και η διευκρίνηση, η εξειδίκευση θα έλεγα, την οποία προσφέρει η τροπολογία 22 για τον έλεγχο του τύπου. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με την 23. Θα πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε ότι μια ετικέτα ποιότητας θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μόνο για τα γεωργικά προϊόντα τα οποία προέρχονται πλήρως από ευρωπαϊκές παραγωγές. Θεωρώ επίσης ότι είναι θετικές οι τροπολογίες 33 και 34 γιατί ακριβώς ασχολούνται με τα οποροκυπευτικά και με την αγορά των οποροκυπευτικών με σωστό τρόπο. Συμφωνώ επίσης με τον κύριο Ταμπάτζη με την τροπολογία 55. Ζητά να υπάρξουν κάποιες διευκρινήσεις για τις βασικές πρώτες ύλε, τα βασικά συστατικά των τροφίμων που έχουν ε, μετασχηματιστεί και για τα οποία η υπάρχουσα κοινοτική νομοθεσία δεν τα αντιμετωπίζει επαρκώς. Σχετικά με τις τροπολογίες 65, 66 και 67, καλώ τους συναδέλφους να εξετάσουν τη σημασία που έχει να υποδεικνύεται ο τόπος παραγωγής ακόμα και στα μετασκευασμένα ή στα επεξεργασμένα προϊόντα. Θεωρώ επίσης ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η διευκρίνηση που γίνεται μέσω της 86, 109 και 112 από τον Δεκάστρης και άλλους όπως επίσης και την 108 της συναδέλφου Γαρσία για την ανάγκη να υπάρχουν περισσότεροι πόροι για τις εκστρατείες προώθησης των προϊόντων και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συμφωνώ και με την 114 της συναδέλφου Γκαρσία. Δεν θα ήθελα να σας καθυστερήσω, θα συμφωνήσω με αρκετούς άλλους συναδέλφους οι οποίοι έχουν κάνει κάποιες συγκεκριμένες διευκρινήσεις με τις τροπολογίες 120 και 128 για την προστασία των προϊόντων μας στα πλαίσια των κανόνων του ΠΟΕ και σχετικά με το σεβασμό των κανόνων που με τη σειρά του σέβονται το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς, θα ξεκινήσει λοιπόν η συζήτηση. Η αποδοχή της έκθεσης αυτής θα γίνει επίσημα στις 22 και 23 Φεβρουαρίου. Έχουμε δηλαδή τον απαιτούμενο χρόνο για να εμβαθύνουμε. Ευχαριστώ τον κύριο Σκοτά. Δίνω το λόγο στον κύριο Χεράνς Γαρσία. Στην κυρία Χεράνς Γαρσία. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν είχα ακριβώς με οργανωμένο τρόπο τις τροπολογίες έτσι όπως τις παρουσίασε ο κύριος Σκοτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σκοτά για την κρίση την οποία εξέφρασε σε σχέση με τις τροπολογίες μου. Στα πλαίσια των έψιλων ε, ε, προφανώς και οι πρωτοβουλίες οι οποίες θα προστατεύσουν τα προϊόντα μας είναι απαραίτητες για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υψηλής ποιότητας. Δεν θα πρέπει επίσης να αγνοήσουμε ότι το σύστημα εγγυήσεων για την ονομασία προέλευσης είναι κάτι το οποίο συνδυάζεται με τα πήγαμα ε εύκολα. Οι πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι πάντα οι καλύτερες σχετικά με τους κανόνες εμπορίας των προϊόντων. Προφανώς και είμαστε υπέρ της δημιουργίας κάποιων ετικετών που να αφορούν αποκλειστικά τα ορεινά λεγόμενα προϊόντα. Θέλει όμως πάρα πολύ μεγάλη προσοχή εδώ η υπόδειξη επίσης κάποιων ειζημάτων ή καταλήπων τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις ετικέτες των προϊόντων των μεταποιημένων τα οποία κυκλοφορούν. Δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι, δεν έχουμε τις μεθόδους που απαιτούνται και πρέπει να είμαστε σοβαροί. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει συγκεκριμένη αναφορά στη λεγόμενη ολοκληρωμένη γεωργική παραγωγή. Η γεωργία αυτή, η γεωργική αυτή δραστηριότητα θα πρέπει να είναι απόλυτα διαφανής για τους καταναλωτές, θα πρέπει να είναι απόλυτα ενήμεροι οι καταναλωτές για τους τρόπους παραγωγής σχετικά με, τα, με την ονομασία συγκεκριμένων προϊόντων, προϊόντων ειδικής ποιότητας. Νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε σε αυτού του είδους τα προϊόντα γιατί έτσι θα βοηθήσουμε τους παραγωγούς. Ατέ. κύριε Περές, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σκοτά για την προσπάθεια την οποία έκανε ε, σε μια έκθεση που παρουσιάζει πάρα πολύ ενδιαφέρον και η οποία αντιμετωπίζεται και αυτό το δείχνουν οι τροπολογίες που έχουν κατατοθεί με πολύ διαφορετικό τρόπο. Πρέπει να κάνω να ξεκινήσω κάνοντας δύο παρατηρήσεις σχετικά με τις ετικέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημερίζομαι το ότι τα μεταποιημένα ή επεξεργασμένα γεωργικά προϊόντα θα πρέπει να μεταποιούνται και να γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό δεν θα πρέπει να δημιουργεί επιπλέον κόστος για τους παραγωγούς. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ζητήσουμε οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε πώς θα λειτουργήσουν τα καθεστώτα αυτά ιδιωτική πιστοποίησης. Πρέπει να συμπληρώνονται από τους αρμόδιους φορείς και να υπάρχει συμφωνία όσον αφορά την προσθέμενη αξία που θα έχουμε τελικά από αυτά τα προϊόντα. Ευχαριστώ. Ο σκιώδης εισηγητής κύριο Σταμπάτζη έχει το λόγο. Ε, Σχετικά με την ομάδα των σοσιαλιστών. Υπάρχει δυνατότητα συνένεση σε τέσσερα θέματα. συμφωνία ανάμεσα στις ε, πολιτικές ομάδες και στην πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής που υποστηρίζουν την ετικέτα προϊόντων ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πι όμικρον πι και πι γάμα ε μπορούμε να δεχθούμε τις προτάσεις του κυρίου Σκότα και επίσης συμφωνούμε και για την οργανική καλλιέργεια να υπάρχουν ειδικέ ετικέτες για προϊόντα που παράγονται από τέτοιου είδους καλλιεργίες και επίσης υπάρχει και δεχόμαστε και η δυνατότητα εθελοντικής ετικετοθεσίας των προϊόντων ορεινών περιοχών. Καταρχάς τώρα ο τόπος παραγωγής. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες οι οποίες αποδεικνύουν ότι ορισμένοι συνάδελφοι δεν έχουν ενημερωθεί σωστά για το ότι τα βασικά προϊόντα, για τα βασικά προϊόντα σήμερα, σήμερα επαναλαμβάνω, είναι υποχρεωτική η αναγραφή του τόπου παραγωγής, σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανονισμούς. Το βασικό θέμα το οποίο, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Σκοτά είναι οι ετικέτες για τα μεταποιημένα προϊόντα. Σχετικά με τα προϊόντα αυτά έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα θα πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά με την υποχρεωτική ετικετοθεσία των μεταποιημένων προϊόντων. Γιατί στην Αυστραλία, στη ΣΥΠΑ, στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού υπάρχει ένα σύστημα ετικετοθεσίας και θα ήταν μειονέκτημα για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έχουν ένα αντίστοιχο σύστημα για τα προϊόντα αυτά τα μεταποιημένα. Θα πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαμορφώσει ένα νέο σύστημα και να ορίζονται σωστά τα βασικά συστατικά. Ο κ. Ντόρφμαν κατέθεσε μια τροπολογία την οποία μπορούμε να υποστηρίξουμε και να καταλήξουμε στο τι σημαίνουν βασικά συστατικά. Δηλαδή ποσοστιαία τι αντιπροσωπεύουν, σε επίπεδο προστιθέμενης αξίας τι αντιπροσωπεύουν. Ε, θυμίζω εδώ ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, στην οποία είμαι αναπληρωτής, δεν υποστηρίζει τις προτάσεις μας και για τα μεταποιημένα προϊόντα και για τα βασικά κυρίαρχα γεωργικά προϊόντα. Σχετικά με τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Γίνεται μεγάλη συζήτηση εδώ γιατί δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για να υπολογιστεί το ίχνος σε άνθρακα. Πιστεύω όμως ότι για να μπορέσουμε να διασώσουμε την πολιτική μας στον τομέα της γεωργίας και τη γεωργία ειδικά θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιο τρόπο μέτρησης του ίχνους παραγωγής άνθρακα για τα γεωργικά προϊόντα και ιδιαίτερα ε, για ε, το ίχνος το λεγόμενο οικολογικό το οποίο αφήνουν τα προϊόντα αυτά. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να δείξουμε την εισφορά της Ευρωπαϊκής Γεωργίας στην προστασία του περιβάλλοντος. Σχετικά τώρα με την εθελοντική ετικετοθεσία για προϊόντα ελεύθερα γενετικά τροποποιημένων ουσιών και προϊόντων, θα πρέπει να βρούμε μία λύση. Εδώ έχουμε ακόμα κάποιες διαφορές έχει σημασία όμως να βρεθεί μια λύση για την πολιτική ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και για να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι η γεωργία μπορεί να συνεισφέρει με αηφόρο τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ κύριε Ταμπάτζη. Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά. Μικρό. Ευχαριστώ. Άκουσα αυτά που είπε και ο συνάδελφο για τις κατευθυντήριες γραμμές που στηρίζουμε στην έκθεση αυτή. Πρόσθεσε επίση και κάτι για τη δουλειά που έκανε ο εισηγητή. Συγχαρητήρια βέβαια. Και πάνω απ' όλα πρέπει να πούμε στο σώμα ότι για το θέμα αυτό πρέπει το μήνυμά μας να είναι πολύ δυνατό όσον αφορά τη συζήτηση που γίνεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Γιατί η χειρότερη απειλή που μπορεί να πέσει πάνω στην πολιτική αυτή που θέλει να προωθήσει την ποιότητα, τη σχέση ε, ανάμεσα στα γεωρικά προϊόντα και το χώρο που παράγονται, είναι η διαπραγματεύσει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Συνεπώ, για τι τροπολογίε που προτείνονται και για τη λογική του εισηγητή, πρέπει να φροντίσουμε να πετύχουμε ευρεία συνένεση προκειμένου να στηρίξουμε τη γραμμή αυτή στα πλαίσια του ΠΟΕ και να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα επ' αυτού στην Κομισιόν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ Στεφάν. Νικουλέσκου, αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στον κύριο Σκότα για το έργο του. Έχω ένα πολύ σύντομο σχόλιο παρακαλώ πιστεύω ότι όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων υπάρχουν διάφορες ενδείξεις, ποιοτικές ενδείξεις. Και δεν είναι ο ένας δείκτης εναλλακτικό με τον άλλον, όχι. Όλες οι ενδείξεις είναι σημαντικές για την ποιότητα. Όλοι οι δείκτες. Η παραγωγή, μην το ξεχνάμε, θέλουν οικονομική στήριξη για να μπορούν να παράγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα. Και εδώ έχουμε το δεύτερο πυλώνα κυρίως. Αλλά αυτό που πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην έκθεση είναι ακριβώς αυτό, γιατί δεν το αναφέρει αυτό αρκετά. Ευχαριστώ κύριε Νικουλέσκο. Ντόρφμαν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προσπάθεια την οποία έχει κάνει Δύο πράγματα θέλω να υπογραμμίσω. Νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε κάθε πρόταση η οποία ερμηνεύει σωστά το σύστημα των προϊόντων αυτών και το ετικετοθεσίας τους. Θα πρέπει το σύνολο του τομέα παραγωγής να αποφασίζει και για το πότε και για το πώς θα προωθήσει εμπορικά τα προϊόντα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί καμιά φορά οι νόμοι αντιτράστ δημιουργούν ορισμένα προβλήματα, τουλάχιστον στη δική μου χώρα. Και θα πρέπει εδώ να δούμε ότι συνήθως τα ωφέλη από τέτοιου είδους εμπορικές προσπάθειες ωφελούν περισσότερο την βιομηχανία και όχι τόσο τους γεωργούς. Είναι θετικό το ότι έχουμε αναφερθεί και στη δυνατότητα ετικετών για προϊόντα ορεινά από ορεινές περιοχές αλλά δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε μία αντίθεση θα έλεγα ανάμεσα στα βιολογικά προϊόντα και στα, και στα προϊόντα pop. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι χαρακτηριστικά με σε διαφορετικά επίπεδα και δεν θα πρέπει να δημιουργείται μια σύγχυση. Τα pop είναι συγκεκριμένα προϊόντα, μπορεί να μην είναι βιολογικά προϊόντα, μπορεί και να είναι, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στα δύο. Ευχαριστώ κύριε Ντόρφαν. Μποβέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον εισηγητή για τη δουλειά του. Ήδη έχει καταλήξει σε μια πολύ καλή σύνθεση. Έχω όμως να προσθέσω κάποια σημεία τα οποία δεν θυγηθήκαν ακόμα. Για παράδειγμα, σαφήνεια, διαφάνεια. Είναι ανάγκη να υπάρχουν όσον αφορά την προέλευση των υλών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα ε, με προέλευση Γιατί όταν μιλάμε για την ποιότητα πρέπει να υπάρχει και έλεγχος των όγκων, των ποσοτήτων που φτάνουν στην αγορά. Και πρέπει να υπάρχει συνοχή ανάμεσα στην ποσότητα που διατίθεται στην αγορά για να δούμε αν η αγορά μπορεί να την απορροφήσει. Έτσι, συγχρόνως, ο παραγωγός μπορεί να ξέρει τι θα βγάλει. Θέλω επίσης να επιμείνω και όσον αφορά την διαχείριση των δικτών ποιότητας. Πρέπει να στηρίξουμε τους οργανισμούς διαχείρισης που βρίσκονται επί τόπου, διότι η ποιότητα πρέπει να ενισχύεται από την τοπική διαχείριση. Είναι σημαντικό λοιπόν τα μέσα αυτά να μπορούν να υπάρχουν και να αναπτύσσονται. Συγχρόνως πρέπει να υπάρχει και οικονομική στήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να στηρίξουμε την διαχείριση αυτή σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο όταν πρόκειται για προϊόντα ονομασία προελεύσεω. Θέλω επίσης να επιμείνω, τελειώνοντας και στην ανάγκη που υπάρχει, τα μέσα λειτουργίας να επιτρέπουν να έχουμε προϊόντα με βιοπικιλότητα. Διότι είναι ποιότητα και αυτή η βιοπικιλότητα. Επίσης, να διατηρήσουμε τη σχέση με μικρές και μεσές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με τη γη, γιατί και αυτό είναι σημείο που δείχνει ποιότητα. Τέλος, πρέπει να επιμείνουμε στη δημιουργία απασχόλησης. Μπορούμε να δημιουργήσουμε απασχόληση άμεσα και έμεσα χάρη σε αυτούς τους δείκτες ποιότητας. Και όπως έλεγα και πριν, η ποιότητα αυτή είναι τεράστια σημασίας στους δύσκολους χώρους για να στηριχθούν οι μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του. Σημείωσα ότι έλαβε υπόψη του την τροπολογία που Πρόεδρε συζητήσαμε και προτείναμε πολύ από εμά όσον αφορά την ποσότητα και τη σημασία που έχει η ποσότητα όγκος του προϊόντος σε σχέση με την ποιότητα. Τώρα για τις παρατηρήσεις που έγιναν. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάμε ακόμα πιο μακριά στην διατήρηση της ταυτότητας του προϊόντος κατά τη διάρκεια ολόκληρης της εμπορικής αλυσίδας. Είναι πολύ σημαντικό οι δομές που σχετίζονται με την γεωγραφική ένδειξη, με την ονομασία προέλευσης, να παρεμβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια της αλυσίδας και στη συσκευασία. Γιατί ακριβώς αυτή είναι μια πρόσθετη αξία και εκεί είναι που κινδυνεύει το προϊόν. Έτσι λοιπόν θέλω και εγώ να πω ότι η μεγάλη σημασία που έχουν τα προϊόντα ποιότητας είναι ότι βοηθούν την τοπική κοινότητα που βρίσκεται σε δυσκολία. Είναι μια πρόσθετη αξία, την οποία δεν πρέπει να την πάρει, να επωφεληθεί από αυτήν κάποιος άλλος ξένος, άσχετος με τον τόπο που παράγεται το προϊόν ποιότητας. Καλώ. η συζήτηση έχει ενδιαφέρον, το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο και θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριος Κορντονιέ. για να κλείσουμε πάλι με τον εισηγητή μας, τον κύριο Σκοτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον εισηγητή, αλλά και όλους όσοι συμμετείχαν στην ε, συζήτηση αυτή, αλλά και με τις τροπολογίες που κατέθεσαν η Επιτροπή, φυσικά και χαίρεται όλος ιδιαιτέρως που υπάρχουν τόσες τροπολογίες στην έκθεση, γιατί αυτό δείχνει πόσο μεγάλο ενδιαφέρον έχετε για αυτό το θέμα. Τώρα επιτρέψτε μου παρακαλώ να κάνω μερικές παρατηρήσεις μόνο. Όσον αφορά το σήμα, το EU, αν πρόκειται για ένα σήμα το οποίο δείχνει την προέλευση των προϊόντων, ότι προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τότε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μελετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό αναφέρεται και στην ανακοίνωση. Όμως, αν πρόκειται για ένα σήμα το οποίο βεβαιώνει ποιότητα, ποιότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει ότι πρέπει να την έχουν όλα τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αυτό δεν προβλέπεται. Τουλάχιστον, σύμφωνα με τις αναλύσεις μας, δεν μπορούμε να προβλέψουμε κάτι τέτοιο για... Μάλλον δεν μπορούμε κάτι τέτοιο να το απαγορεύσουμε εφόσον το ε, καταστήσουμε ε, θεσμό από προϊόντα που έρχονται από τρίτες χώρες που σέβονται τις ίδιες προδιαγραφές. Τώρα, όσον αφορά την προέλευση του προϊόντος, δεν ξέρω αν σας κατάλαβα καλά, αλλά έχω την εντύπωση ότι είπατε ότι είναι ήδη για τα πρωτογενή προϊόντα ήδη, για τις πρώτες ύλες δηλαδή, ήδη ισχύει, ότι είναι ήδη υποχρεωτικό. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί υπάρχουν κάποια προϊόντα σήμερα για τα οποία δεν υπάρχει τέτοια απέτηση. Για παράδειγμα χείριο κρέας. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε εμείς ότι καλό θα ήταν να μελετηθεί περισσότερο σε βάθος αυτό το ζήτημα. Κάτι ακόμα. Η παρατήρηση που έγινε για τον ΠΟΕ και όσον αφορά τη γεωγραφική ένδειξη. Υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση, αλλά είναι προφανές ότι αποτελεί μέρος των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής <coughs> Επιτροπής της διαπραγματεύσεις που κάνει με τον ε, ΠΟΕ και στα πλαίσια του γύρου της Δόχα. Προφανώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αναγνωριστεί αυτό το σύστημα ποιότητας από τους εμπορικούς μας εταίρους. Και δύο ακόμα σημεία για τα ορεινά προϊόντα. Βέβαια, χαιρόμαστε που βλέπουμε να υπάρχει στήριξη των Ευρωβουλευτών για αυτή την ιδέα. Καλύτερα δηλαδή να εντοπίζονται τα ορεινά προϊόντα προέλευσης απορρινούς χώρους. Θα γίνει μια μελέτη, έχει ήδη ξεκινήσει μάλιστα, για να μελετήσουμε κατά πόσο αυτό είναι εφικτό και τι αποτελέσματα θα έχει. Τέλος, για τη διαχείριση των ποσοτήτων. Θα υπάρξει μια έκθεση, γιατί το Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Health Check να κάνουμε λοιπόν έκθεση όσον αφορά τις ε, γαλακτοκομικές ποσοστώσεις και την ε, προέλευση των προϊόντων αυτών. Την έκθεση αυτή θα τη δώσουμε μέχρι το 2012, αν δεν απατώμε. Και έτσι θα δούμε κάπως πώς επηρεάζονται τα προϊόντα με ονομασία προέλευσης από μια τέτοια διαχείριση. Στα πλαίσια των γεωργικών ε, ενδείξεων, ε, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει περιορισμό του αριθμού των παραγωγών που θα μπορούσαν να αποφεληθούν από την ε, γεωγραφική ένδειξη εφόσον όντως σέβονται την απαιτούμενη ποιότητα. Αυτά, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για άλλη μια φορά λέω, χαίρεται που μπορεί να έχει διάλογο με την Επιτροπή σας. Μάλιστα, κυρίως επειδή σήμερα ξεκινάει η συνθήκη της Λισαβόνας, οπότε εφ' εξής, θα συνεργαζόμαστε όλο και περισσότερο μαζί σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το γνωρίζουμε αυτό και το έχουμε υπενθυμίσει εξ αρχής. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δίνω το λόγο στον κύριο Σκοτά υπενθυμίζοντας σε όλους ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε τις τροπολογίες αυτές και να υιοθετήσουμε το ψήφισμα αυτό στις 22 και 23 Φεβρουαρίου του 2010. Έχουμε κάποιο χρόνο λοιπόν για να σκεφτούμε μέχρι τότε. Τζακάβλο Σκοτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Με τη δική σας βοήθεια Νομίζω έχουμε σχετικά προχωρήσει στα πλαίσια αυτής της έκθεσης. Θα κλείσω με μια σκέψη η οποία θα μου άρεσε πολύ θα έλεγα. Να δω τους παραγωγούς οι οποίοι ασχολούνται με την καλλιέργεια και με τη μεταποίηση των προϊόντων να επιβραβεύονται από τον καταναλωτή ο οποίος επιλέγει το προϊόν τους. Αυτό νομίζω είναι ο βασικός στόχος όλης αυτής της συζήτησης που κάνουμε μέχρι τώρα. Αυτός που δουλεύει, αυτός που υδρώνει και αυτός που δεν κερδίζει, γιατί ξέρουμε ότι η κατανάλωση κάποιων προϊόντων ευρωπαϊκών γεωργικών έχει αρχίσει να πέφτει τα τελευταία χρόνια, είναι κάτι το πάρα πολύ αρνητικό. Ενώ αντίθετα θα πρέπει ο καταναλωτής να μπορεί να καταναλώσει επιλέγοντας και να μην αποφασίζει γι' αυτόν κάποιος άλλος. Καλώς ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Τζακάβλο Σκοτά και περνάμε στο επόμενο σημείο της ενημερήσιας διάταξης, το 6. Relazione libro verde della Commissione sulla gestione dei... Πράσινη βίβλος για τη διαχείριση των των βιολογικών αποβλήτων. Ξέρετε ότι η πράσινη βίβλος της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών προϊόντων έχει σαν στόχο την κοινή δράση. Συνδυασμό των προσπαθειών για τη διαχείριση της αντιμετώπισης των βιολογικών αποβλήτων, ιδιαίτερα των πράσινων αποβλήτων που προέρχονται από κήπους, από καλλιέργειες αλλά και από την κουζίνα των οικειών. Δίνω το λόγο στον Σαλβατόρε Καρόνα, για να παρουσιάσει την έκθεσή του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Πράσινης Βίβλου έχει προωθήσει κάποιες σκέψεις και κάποια συζήτηση για την ανάγκη που υπάρχει να αναλυφθεί μια κοινή κοινοτική δράση σχετικά με τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων διοδιασπόμενων αποβλήτων. Υπάρχει μια συνεχώς μεγαλύτερη παραγωγή αποβλήτων με πολύ μεγάλη απώλεια ενέργειας και με αυξανόμενες περιβαλλοντικές βλάβες στο περιβάλλον και στην υγεία. Συνεπώς, θα πρέπει αυτές οι αρνητικές πλευρές να μειωθούν. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί μια κοινωνία ανακύκλωσης η οποία να χρησιμοποιεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τους πόρους που έχει στη διάθεσή της. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν ο τομέας των οργανικών αποβλήτων, των βιοδιασπόμενων οργανικών αποβλήτων προσφέρει αρκετά μεγάλο χώρο βελτίωσης της κατάστασης της διαχείρισης αυτής για τα οργανικά βιοδιασπόμενα προϊόντα σε επίπεδο κανονισμών, αν θα έλεγα, βρισκόμαστε σε μια αρχική φάση. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη. Για να σας δώσω μια ιδέα για το τι συζητάμε σε επίπεδο ποσοτικό, στην ουσία αναφερόμαστε στο 1 τρίτο περίπου των αστικών αποβλήτων 200.000 τόνους τροφίμων όπως επίσης και αποβλήτων από κήπους, 37 εκατομμύρια τόνους από την βιομηχανία τροφίμων και τη βιομηχανία ποτών που παράγονται ε, μέσα σε ένα χρόνο. Χωρίς να υπάρξει λοιπόν μια αποτελεσματική ανάλυση δράσης και μιας και τα προϊόντα αυτά μπορούν να μεταποιηθούν, να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας και να παράγουν ενέργεια, χάνουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Όπως επίσης περιγράφεται στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μια συγκεκριμένη σειρά προτεραιοτήτων. Πρώτον, να προωθήσουμε την πρόληψη. Δεύτερον, να ενισχύσουμε την ανακύκλωση. Τρίτον, να ευνοήσουμε την συλλογή και την ανάκτηση των προϊόντων αυτών για ενεργειακούς λόγους, για παραγωγή ενέργειας δηλαδή, και μόνο σαν τελευταία επιλογή να χρησιμοποιήσουμε τις χωματερές. Αυτή η επιλογή είναι η λιγότερο επιθυμητή διότι παράγεται θα έλεγα παράγονται και λίματα τα οποία μπαίνουν στους υδάτινους ορίζοντες υπάρχει και παραγωγή φυσικού αερίου ή μάλλον ε, ε, διοξιδίου του άνθρακα ε, που μολύνει και την ατμόσφαιρα. Υπάρχει μια διπλή μόλυνση λοιπόν και πρέπει να το αποφύγουμε και να ευνοήσουμε άλλες επιλογές κυρίως την της ανακύκλωσης μέσω της βιολογικής επεξεργασίας, τα λεγόμενα κόμποστ και επίσης και την καύση αλλά μόνο με ανάκτηση υψηλού ποσοστού ενέργειας. Δεν θα μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μια επιλογή, επιτροπή συγγνώμη, σαν την δική μας, αντίθετα από αυτό το οποίο γίνεται σήμερα στις χωματερές, να προτείνει λύσεις για τον σεβασμό της γης, του εδάφους και των υδάτων όπως και της ατμόσφαιρας. Βλέπουμε ότι στο εσωτερικό των κρατών μελών υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην χρήση των διαφόρων επιλογών. Υπάρχει έτσι λοιπόν ο κίνδυνος μεσοπρόθεσμα να δημιουργηθούν και να παγιωθούν καταστάσεις διαφορετικές με αρνητικές επιπτώσεις και σε περιβαλλοντικό αλλά και σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Γνώμη μου λοιπόν είναι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ακόμα δεν έχει εγκατασταθεί, να αξιολογήσει με την απαιτούμενη δέουσα προσοχή την κατάσταση και να θέσει συγκεκριμένους κοινού μετρήσιμους στόχους για την διαφοροποιημένη συλλογή των αποβλήτων και απορριμμάτων, να υπάρξουν συγκεκριμένες παράμετροι ποιοτικέ και για το κομπόστο και θα πρέπει να υπάρξει σεβασμός γενικότερα και στις αγροτικές γέες στην Ήπεθρο. Αυτές είναι οι προτεραιότητες. Και παράλληλα με όλα αυτά είναι απαραίτητο να ευνοήσουμε και την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών ικανών να συνεισφέρουν στον στόχο μείωσης της μόλυνσης του περιβάλλοντος και να πετύχουμε αυτό το 20% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2020. Να προωθήσουμε επίσης και μέσω μιας πιο εντατικής και αποφασιστικής χρήσης του φορολογικού μέσου να προωθήσουμε έλεγα συστήματα διαφοροποιημένης συλλογής στην πηγή παραγωγής. Συνεπώς η πράσινη βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια εξαιρετική βάση συζήτησης για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πολύ σημαντική θεματολογία της διαχείρισης των βιοδιασπόμενων βιολογικών αποβλήτων. Θα πρέπει να στραφούμε στην ανάγκη να μειώσουμε μέσω ακριβώς και του καθορισμού συγκεκριμένων μετρήσιμων κοινών στόχων. Να μειώσουμε τις διαφορές που ισχύουν ανάμεσα στα διάφορα κράτη. Υπάρχουν χώρες σαν παράδειγμα οι οποίες χρησιμοποιούν την καύση και έχουν υψηλά μερικές φορές επίπεδα ανάκτησης ενεργειακής Γαλλία, Δανία και τα λοιπά Άλλες χώρες όπως η Γερμανία και η Αυστρία αναπτύσσουν δικές τους πολύ μεγάλες δυνατότητες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας προϊόντων για παραγωγή κομπόστ και άλλες χώρες, ιδιαίτερα οι νέες χώρες, υπάρχει πολύ μεγάλη χρήση των χωματερών. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε κάπως τα πράγματα να τα φέρουμε σε μια ισορροπία και η συζήτηση η οποία θα πρέπει να γίνει και εδώ ευχαριστώ τους συναδέλφους που έχουν συνεισφέρει ήδη πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποιες λύσεις. Ευχαριστώ κύριε Καρόνα. Σε αυτή την φάση ανοίγει η συζήτηση. Έχει ζητήσει το λόγο ο Μάρκ Ταραμπελά. Ευχαριστώ. Δύο παρατήσεις έχω να κάνω. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για τις καλές πληροφορίες που μας δίνει για το τι γίνεται στην Ευρώπη. Τώρα για την επιλογή, ε, την κατανομή των σκουπιδιών, όντω σε ορισμένες χώρε. Ε, έχει προχωρήσει πάρα πολύ γιατί τα ανακυκλούμενα είναι χωριστά, τα μέταλλα είναι χωριστά, τα εφάσματα. Οπότε τελικά τι μένει μένει ο σκουδοντενικές μέσα στον οποίο βάζουμε όλα τα υπόλοιπα. Και όλα τα υπόλοιπα είναι τελικά 40% ε, προϊόντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οπότε εμείς από 1η Απριλίου μέσα από ατομικούς κάδους που μπορεί να είναι και 40 λίτρων μαζεύουμε χωριστά τα οργανικά απόβλητα. Και τι διαπιστώνουμε, διαπιστώνουμε ότι τελικά αυτά που πάνε στην καύση είναι 40%. Συνεπώς υπάρχει ακόμα περιθώριο και γι' αυτό θέλω να ενθαρρύνω να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή γιατί μπορούμε πραγματικά τα βιολογικά απόβλητα να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα πηγαίνουμε για καύση. Τώρα εγώ δεν κοιτάω πολύ τηλεόραση αλλά κατά σύμπτωση χτες έπεσα πάνω σε ένα ρεπορτάζ της γαλλικής τηλεόρασης που ήταν για τα απόβλητα των φούρνων. Κοιτάξτε, εγώ είμαι πολύ τυχερός, ποτέ δεν πίνασα στη ζωή μου. Οι γονεί μου, οι παππούδες μου όμως πίνασαν. Και δεν πετάμε το φαγητό, έτσι έχω μάθει. Το ψωμί, το ξερό, το δίνουμε στα πουλιά. Δεν το πετάμε όμως ποτέ στο τενεκέ. Ίσως λοιπόν πρέπει να επιμείνουμε λιγάκι πάνω στο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Γίνεται σε ορισμένου χώρου. ας πούμε ε, το αλεύρι που μας περισσεύει, τι το κάνουμε, το δίνουμε για ζωοτροφές. Δηλαδή να φροντίσουμε να περιορίσουμε τα απόβλητα της βιομηχανία τροφίμων για να μην καταλήγει στο σκουπίδο αλλά να χρησιμοποιείται. Μπορεί να είναι για τα ζώα, εντάξει, ακόμα καλύτερα αν είναι για τους ανθρώπους, γιατί ορισμένοι τρώνε μπαγιάτικο ψωμί, δεν θέλουν μόνο φρέσκο. Είναι και αυτό κάτι πάνω στο οποίο θα μπορούσαμε να επιμείνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, κύριε Δήμεση, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Καρόνα για την ενδιαφέρουσα επισκόπηση της έκθεσης που έδωσε. Είμαι υπέρ του να διεξαχθεί μια σε βάθος συζήτηση του θέματος, διότι άλλωστε έχουμε και πολλά νομοθετήματα που αναφέρονται στο θέμα αυτό, γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα να μην προκαλέσουμε και άλλη περαιτέρω γραφειοκρατία. Ίσως καλύτερα είναι να συνοψίσουμε ορισμένα νομοθετήματα, να τα συγχωνεύσουμε αν θέλετε, ώστε να γίνουν πιο εύληπτα. Σε ό,τι αφορά την επικουρικότητα, να φροντίσουμε ώστε να επιτρέψουμε αρκετή ελευθερία ελιγμών στις περιφέρειες και ένα άλλο πράγμα που θεωρώ ότι είναι σκόπιμο, να καθοριστούν ορισμένα κριτήρια για το πώς ποια μεταχείριση θα υποστούν τα διάφορα αυτά βιολογικά κατάλοιπα, ώστε να έχουμε, να θεσπίσουμε μια μεταχείριση τέτοια που να μπορεί να επιτρέψει για παράδειγμα τη χρήση τους ως λοιπασμάτων στη γεωργία. Είναι τέτοια μορφής και ποιότητας που να μην υπάρχει πρόβλημα να χρησιμοποιηθούν για τους λόγους αυτούς. Μακίνηση. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη για την προσέλευσή μου με κάποια καθυστέρηση. Ευχαριστώ τον κύριο Καρόνα. Η Επιτροπή Αναφορών είχε ένα θέμα γεωργικό ένα θέμα γεωργικό στην ημερήσια διάταξή της, την επισήμανση των προβάτων, δηλαδή με ε, ειδικέ ετικέτες. Εάν χρησιμοποιηθούν τα βιολογικά αυτά απορρίμματα ως ε, λιπάσματα, χρειάζεται πολύ αυστηρή έλεγχη ποιότητας, διότι Καμιά φορά κάποιε πρακτικές που τι θεωρούμε ικανοποιητικέ προκαλούν ωστόσο στο τέλος προβλήματα. Ορισμένα για τα πράγματα που είπε ο κ. Σταραμπέλα και με τα οποία είμαι σύμφωνη γιατί πετιούνται στα σκουπίδια πολλά τρόφιμα. Θα θυμάστε όμως και πέρσι στην Ιρλανδία που είχε υπάρξει ένα πρόβλημα διοξίνη. Πρέπει και εκεί λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι ανακυκλώνουμε και με ποιο τρόπο τα ανακυκλώνουμε. Χρειάζονται και εδώ αυστηρή ποιοτική έλεγχη, διότι καμιά φορά δεν μπορούμε να προβλέψουμε όλα τα ενδεχόμενα προβλήματα. Γι' αυτό όσο πιο προσεκτικοί είμαστε τόσο καλύτερα. Στο πρακτικό επίπεδο οι αγρότες θα προτιμούσαν να υπάρχει περισσότερη συνεκτικότητα σε ό,τι αφορά την μεταχείριση των βιολογικών αποβλήτων. Πρέπει να κατανοήσει και το κοινό ότι εάν θέλουν να ανακυκλώνουν και να κάνουν και το λεγόμενο compost, να επιτρέπουν τη σήμωση αυτή δηλαδή που επιτρέπει στο τέλος να γίνονται χρήσιμα τα πράγματα αυτά για λοιπάσματα κτλ. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί καμιά φορά τα αποτελέσματα είναι απρόβλεπτα. Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν ποιες είναι οι ενδεχόμενες αυτές οι επιπτώσεις. Θα συμφωνήσω με την ιδέα που είπαν ορισμένοι προηγούμενοι συνάδελφοι ότι ίσως χρειάζεται να συνοψιστούν κάποια νομοθετήματα, διότι έχουμε αρκετούς κανόνες, αλλά δεν γίνεται συντονισμό τους, είτε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε και στο εθνικό. Θα συνεχίσουμε. Housing. Είναι σωστό ότι έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ διαφορετικές προδιαγραφές αναχώρα και για τον χωρισμό των απορριμμάτων αλλά και για τη χρήση τους για παραγωγή ενέργειας. Τώρα, το να διαχωρίζονται τα απορρίμματα και στο τέλος να καταλήγουν σε καύση, ούτε και αυτό είναι σκόπιμο. Εγώ νομίζω ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλά με σωστό τρόπο για την δημιουργία βιολογικού αερίου. Μεθανίου για παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να κλείσουν οι κύκλοι. Δηλαδή τα προϊόντα αυτά τα οποία ξεκινάνε από την γεωργική παραγωγή να ξανακαταλήξουν εκεί. Διότι πολύ συχνά καταλήγουν στις εγκαταστάσεις καύσεως, καίγονται και στην ουσία δηλαδή γίνονται αέρια που επιβαρύνουν τον ατμοσφαιρικό αέρα. Gladfelder. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα. Και ιδίω διότι υπάρχουν ε, σοβαρές προβλέψεις που λένε ότι στις επόμενες δεκαετίες θα αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά και δύσκολα προβλήματα και σημαντικά ελλείμματα και στα τρόφιμα και στην ενέργεια. Πρέπει να δούμε πρώτα οι, ποιες είναι οι φυστάμενες ρυθμίσεις στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιες από τις ρυθμίσεις αυτές είναι χρήσιμες να διατηρηθούν. Έχω ήδη συναντηθεί με γεωργούς και άλλους αγρότες που μου είπαν ότι λόγω των ε, περιορισμών που επιβάλλουν η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ορισμένα απορρίμματα για κτηνοτροφές, που θα ήταν το καλύτερο. Γιατί αυτό θα απέδιδε και το περισσότερο, τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Απορρίμματα των μαγειρίων, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθούν για ζωοτροφές. Αυτό σημαίνει, αν χρησιμοποιηθούν εκεί δηλαδή, ότι δεν χρειάζεται να καταλήξουν στα κομπόστ, ούτε να καταλήξουν στην καύση το ερώτημα, για παράδειγμα, ποιες είναι οι νομοθετικές ρυθμίσεις που υπάρχουν που είναι περιτές και οι οποίες μάλλον εμποδίζουν τις περαιτέρω εξέλιξεις. Και αυτό πρέπει να εξεταστεί. Σας ευχαριστώ. Ο Λεύνητσακ και ζητώ συγγνώμη αν δεν προφέρω καλά το όνομά σας. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Καρόνα ιδιαίτερα, τον εισηγητή, ο οποίος ε, ανέπτυξε με ιδιαίτερα λεπτομερό το θέμα. Ασφαλώ και υπάρχουν δυσκολίε με τα απόβλητα και ιδιαίτερα σε ορισμένες χώρες μέλη που αντιμετωπίζουν αρκετά μεγάλα προβλήματα. Δεν θα επαναλάβω τα επιχειρήματα που ήδη ακούστηκαν. Ωστόσο, θέλω να, θέλω να τονίσω την εκπαίδευση του κοινού. Αυτοί που παράγουν τα απορρίμματα, τα απόβλητα, θα πρέπει να μάθουν και να τα χωρίζουν. Εδώ χρειάζεται εκπαίδευση του κοινού σε όλες τις χώρες μέλη. Όταν μιλούμε για βιολογικά απόβλητα και ιδιαίτερα την διαχείριση των αποβλήτων της αγροτικής παραγωγής, εκεί χρειάζεται πραγματικά να κάνουμε μια πάρα πολύ σοβαρή προσέγγιση για την εκπαίδευση των αγροτών. Το τι κάνει ο αγρότης τα απόβλητα της παραγωγής του. Αυτό χρειάζεται πάρα πάρα πολύ δουλειά ακόμη. Νομίζω ότι μίλησαν όλοι όσοι ήταν γραμμένοι στον κατάλογο των ομιλητών. Επιτρέψτε μου και εμένα να κάνω παρακαλώ ένα σχόλιο. Συμφωνώ με τις ανησυχίες σας όσον αφορά τον κίνδυνο υπερβολικής γραφειοκρατίας σε αυτό το τομέα. Ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρακαλώ τώρα. Um, Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο και θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Κορώνα για την τόσο καλή παρουσίαση που έκανε της ε, Πράσινης Βίβλου. Τα σχόλιά του είναι πολύ σωστά. Δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2008 και έχουμε σχόλια ήδη από πολλούς φορείς. Υπάρχει στην ιστοσελίδα η πράσινη βίβλος, οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να την κοιτάξει εκεί. Ε, ουσιαστικά οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι εξέφρασαν λίγο πολύ τις ίδιες ανησυχίες που εκφράσατε και εσείς όσον αφορά την αύξηση της πρόληψης, ώστε να μην έχουμε πολλά απόβλητα από τα τρόφιμα, ε, μήπως μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα επεξεργαστούμε διαφορετικά επίσης και ότι χρειάζεται επίσης και έρευνα για νέες τεχνολογίες που θα μείωναν τα απόβλητα. Τώρα σημειώνω εγώ βέβαια ότι η Επιτροπή σας εξέφρασε διάφορα σημεία τα οποία θα εξεταστούν και στην ε, έκθεση αξιολόγησης ότι χρειάζεται να δούμε καλύτερα το θέμα των βιολογικών αποβλήτων και πώς μπορούμε να μειώσουμε τα απόβλητα αυτά, είτε μέσω καύσης, είτε μέσω ε, ζύμωσης ε, του κόμποστ. Και επίσης πρέπει να δούμε και τις προδιαγραφές. Τι προδιαγραφές υπάρχουν στην κάθε περίπτωση και για ποιο είδος αποβλήτων. Και επίσης να φροντίσουμε να υπάρχει έλεγχος των υλικών που επαναχρησιμοποιούνται. Σημείωσε επίσης ότι η Επιτροπή σας θέλει να δούμε περισσότερο τι γίνεται με την υπάρχουσα νομοθεσία, πριν φτιάξουμε καινούργια δηλαδή. Και να δούμε τι ισχύει στις διάφορες χώρες όσον αφορά την διαχείριση των αποβλήτων. Επίσης, τι θα κάνουμε τώρα στη συνέχεια για αυτό το θέμα. Ολοκληρώνεται η έκθεση αντικτύπου, όπου εξετάζονται όλες αυτές οι αναλλακτικέ και ελπίζουμε να έχουμε μία απάντηση για το προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάμε και πώς. Κοιτάμε και την νομοθετική οδό, αλλά και του ήπιου δικαίου, όπως λέγεται, για να δούμε τι μέσα τελικά θα χρησιμοποιήσουμε. Η Επιτροπή έχει υιοθετήσει τα συμπεράσματά του για αυτή την πράσινη βίβλο ήδη τον Ιούνιο. Οπότε είναι ενδιαφέρον να το ξέρετε αυτό. Εμείς αρχές του 2010 θα ολοκληρώσουμε την έκθεση αντικτύπου μας. Και έτσι πια θα είναι ξεκάθαρο ποια είναι τα συμπεράσματά μας και τι δρόμο θα ακολουθήσουμε από εκεί και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το λόγο έχει τώρα ο συγητής. Παρακαλώ, για να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Παρακαλώ κύριε Σιγητά. Μου φαίνεται ότι η συζήτηση την οποία κάναμε μέχρι τώρα δείχνει ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους. Και υπό το φως των παρατηρήσεων της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομίζω ότι μπορούμε πολλά να προσφέρουμε στη συζήτηση. Ευχαριστώ τους συναδέλφους λοιπόν και θα λάβω υπόψη μου αυτά τα οποία είπατε. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Θα περάσω στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Είναι ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, η οποία είναι υπεύθυνη επί της ουσίας αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας, αποφάσισε να εφαρμόσει το άρθρο 195,5 του κανονισμού και να ζητήσει από την κυρία Σόμερ να παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο και θα πρέπει λοιπόν και η δική μας Επιτροπή να εκφραστεί σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Ο δικός μας εισηγητής είναι ο κύριος Μάρκ Ταραμπελά, ο οποίος εργάστηκε επί τη βάση της πρώτης έκθεσης του Φεβρουαρίου του 2009 της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη και νέες προβλέψεις ε, όπως ε, οι ονομασίες προέλευσης. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον Μάρκ Ταραμπελά για να θυμίσει σε όλους ότι η προθεσμία κατάθεσης των τροπολογιών είναι η 8η Δεκεμβρίου. Η 8η Δεκεμβρίου λοιπόν και η ψηφοφορία θα γίνει στις 27 Ιανουαρίου. Ταραμπελά, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πραγματι, όπως το είπατε, βασίστηκα στην έκθεση που ήδη υπήρχε, που ήδη είχε ετοιμάσει η συνάδελφος Κόρτα το Μάρτιο του 2009. Ε, η διαδικασία όμως ξανάρχισε λοιπόν, οπότε ναι, μεν βασίστηκα σε αυτή την έκθεση γιατί η συγκήτρια είχε κάνει ήδη πολλή δουλειά και οι συνάδελφοι οι οποίοι είχαν προτείνει τροπολογίες, οπότε χρησιμοποίησα όλα αυτά τα στοιχεία και εκτίμησα πάρα πολύ την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν βέβαια διάφορε λεπτομέρειε με τι οποίες δεν συμφωνώ και το λέω. Και χρησιμοποίησα, συμπεριέλευα πολλές ιδέες λοιπόν από την αρχική έκθεση και από τις τροπολογίες των συναδέρφων, ΕΛΚΑ, ΑΛΔΕ, Πρασίνων και άλλων και άλλων. Αυτά. Λοιπόν, να σα πω τώρα τι προτείνω σε έξι σημεία. Πρώτο, σε σχέση με τις πληροφορίες, τις υποχρεωτικές πληροφορίες. Στο Στρασβούργο είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με διάφορους σκιώδεις εισηγητές για να διευκρινίσουμε διάφορα πράγματα. Και βέβαια ξεκίνησε μια ευρύτερη συζήτηση, εννοείται. Λοιπόν, υποχρεωτικές πληροφορίες, λέμε για τα τρόφιμα. Είναι ενδιαφέρον πραγματικά να μπορούμε να προσθέσουμε εδώ κάτι παραπάνω που να δείχνει ποια είναι η χώρα προέλευσης. Για μένα προέλευση και καταγωγή είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Διότι εμένα δεν με ενδιαφέρει το τελευταίο σημείο από όπου ήρθε το προϊόν. Με ενδιαφέρει η πραγματική καταγωγή του, η αρχική του, το αρχικό του σημείο. Αν είναι ένα ζώο ας πούμε που εσφάγει να ξέρω πού. Γι' αυτό κάνω εγώ αυτή τη διάκριση. Άλλο η προέλευση και άλλο η καταγωγή για μένα. Είμαστε στην Επιτροπή Γεωργίας, οπότε έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία για τους παραγωγείς και για την παραγωγή. Υπάρχει μια ολόκληρη αλυσίδα. Ξεκινάμε από τον παραγωγό, φτάνουμε στον καταναλωτή. Υπάρχει ο παραγωγός, υπάρχει ο μεταπητής, αυτοί που χρησιμοποιούν δηλαδή αυτό το προϊόν και υπάρχουν και εκείνοι που το διανέμουν. Γι' αυτό λοιπόν θέλω ο καταναλωτής να μπορεί να ξέρει. Όλοι μιλάμε για τη θέρμανση του πλανήτη. Το είπα και στο Στρασβούργο. Μα δεν είναι μόνο η βιομηχανία, δεν είναι μόνο οι μεταφορές, είναι και η γεωργία που μπορεί να παίξει ένα ρόλο και η κατανάλωση. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι στο μέλλον πρέπει οι καταναλωτές να είναι πιο ενημερωμένοι και να μπορούν καλύτερα να προσέξουν την προέλευση του προϊόντος το οποίο τρώνε. Αν είναι ένα μήλο, ας το έχουμε από μια περιοχή κοντά μας και όχι να αγοράσουμε ένα μήλο το οποίο μας έρχεται από την άλλη άκρη του πλανήτη. Εδώ έχει σημασία να γνωρίζουμε ποιο είναι το πρωταρχικό συστατικό. Εντάξει, δεν θέλω εδώ να βάλουμε παραπάνω γραφειοκρατία. Σε μια ντομάτα μπορεί να υπάρχει αλάτι, μπορεί να υπάρχει και πιπέρι, αλλά υπάρχει ντομάτα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρωταρχικό συστατικό που μας ενδιαφέρει να ξέρουμε την προέλευσή του. Θα ήθελα επίσης και τη διεύθυνση και το όνομα του παραγωγού. Ξέρω ότι δεν γίνεται πάντα, αλλά είναι ενδιαφέρον για ορισμένα τρόφιμα. Και αυτό, αυτό σημαίνει συγγνώμη, ότι υπάρχει και μεγαλύτερο σεβασμό απέναντι στο προϊόν όταν ξέρουμε ότι προχωράει στην αλυσίδα με το όνομά μας και τη διεύθυνσή μας. Έπειτα η παρουσίαση. Εδώ διαφωνώ με την Επιτροπή όσον αφορά το μέγεθος. Τα 3 μιλιμέτρα για μένα δεν λέει τίποτα. Και για πολλά προϊόντα σε μικρές συσκευασίες, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συσκευασία. Και είδαμε τι μελετήσαμε με την προηγούμενη έκθεση. Δεν θέλουμε παραπάνω απόβλητα, λιγότερα θέλουμε. Γι' αυτό νομίζω ότι ένα μιλιμέτρα για τις συσκευασίες ε, ή δύο μιλιμέτρα να έχουμε πάνω από 100 τετραγωνικά εκατοστά είναι ένας καλός συμβιβασμός. Και επίσης είναι απαραίτητο να υπάρχει σημαντική αντίθεση μεταξύ γραμματοσυρών, κοιτάξτε, πήρα κάτι τελευταία, ε, ήταν το φόντο πολύ σκούρο, τα, τα γράμματα πάνω επίσης, ε, πώς να καταλάβω τι λέει εκεί. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει σημαντική αντίθεση. Άσπρο μαύρο ή τέλος πάντων ανοιχτό χρώμα το ένα, σκούρο χρώμα το άλλο, τα γράμματα και ο φόντος, για να μπορούμε να διαβάσουμε καλά τις πληροφορίες έπειτα να είναι τυπωμένες σε μία λία επιφάνεια. Γιατί ο καφές, για παράδειγμα, όταν έχει αφαιρεθεί ο αέρας, καταλήγει με μια επιφάνεια που δεν είναι λία. Άντε λοιπόν να διαβάσεις τι λέει μια επιφάνεια η οποία δεν είναι λία. Δεν γίνεται. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες πρέπει να παρουσιάζονται έτσι που να μπορεί ο καταναλωτής να τις διαβάσει. Υπάρχουν προγράμματα για να χρησιμοποιούμε τις νέες ε, τεχνολογίες για τις μη υποχρεωτικές πληροφορίες. Εντάξει, όλοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ σημεία και πρέπει να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει εκεί και να βλέπει τις υπόλοιπες πληροφορίες, αυτές που δεν είναι υποχρεωτικές δηλαδή. Δεν είμαι κατά, καφέ άλλο. Ε, τώρα, η σαφήνεια των επισημάνσεων για πράγματα τα οποία δείχνουν ε, τη δημιουργική χολυστερίνη για παράδειγμα. Εγώ δεν είμαι μεν επιστήμονας αλλά έχω καθίσει και έχω διαβάσει για τα κορεσμένα, τα κόρεστα. Αλλά υπάρχουν ε, και... Ε, και ουσίες οι οποίες δημιουργούν τρανσαμινικά οξέα που ορισμένοι δεν τα έχουν ακούσει ποτέ στη ζωή τους. Αλλά όλα αυτά πρέπει να δίνονται Ω πληροφορία στον καταναλωτή. Τι δεν έχει ζάχαρη για παράδειγμα από τα προϊόντα. Τι αντίθετα ποιο προϊόν έχει επιπλέον ζάχαρη. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι η φυσική ζάχαρη δεν γίνεται εύκολα λίγο, δεν είναι απορροφά. Ενώ στην αντίθετη περίπτωση όταν δεν είναι φυσική η ζάχαρη δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην υγεία πρέπει υποχρεωτικά να ξέρουμε το καθαρό βάρος. Αν αγοράζουμε 200 γραμμάρια πρέπει να ξέρουμε τι είναι. Είναι μία μονάδα βάρους που είναι κατανοητή και πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται το καθαρό βάρος του προϊόντος. Ε, είπαμε επίσης μήπως είναι καλό να βάζουμε αναμερίδα προσυσκευασμένη. Ναι, αλλά όταν είναι ίσες αξίες μεταξύ τους. Δηλαδή όταν λέμε μερίδα, εντάξει, μερίδα όταν λέμε πάνω στα chips τι σημαίνει. 170 γραμμάρια είναι το πακέτο και τι λέει η βιομηχανία, ναι, 125 γραμμάρια είναι η μερίδα. Και άρα εκεί θα πω πόσες, καλο... πόσες ε, θερμίδες έχει. Ε, ναι, αλλά το πακέτο είναι πακέτο. Οπότε τελικά ο καταναλωτής πολύ δύσκολα φτάνει να υποθέσει ότι αφού η μερίδα είναι 125, αυτό που διαβάζω εδώ για τις θερμίδες αφορά τα 125 γραμμάρια και όχι ολόκληρο το πακέτο. Τι και τα μπισκότα. Όταν δεν είναι συσκευασμένα αναμερίδα, ε, ε, πώς να το υπολογίσουμε αυτό. Όχι, να είναι συσκευασμένα σε μερίδα. Και έτσι να ξέρουμε ότι 100 γραμμάρια είναι η μονάδα αυτή που θέλουμε να ονομάζουμε μερίδα. Στον κανόνα αυτό βάζω μία εξαίρεση που μιλάω για αναλογία. Όταν πρόκειται για κάτω από 100 γραμμάρια, προκειμένου δηλαδή ε, να παρέχεται έγκυρη ενημέρωση. Όταν ένα τρόφιμο ζυγείς λιγότερο από 100 γραμμάρια, η διατροφική δήλωση μπορεί να εδράζεται αποκλειστικά σε μερίδες ή σε μονάδες εάν το τρόφιμο είναι προσυσκευασμένο σε μερίδες ή σε εξατομικευμένες μονάδες ίσες μεταξύ τους. Ε, κοιτάξτε, ένα μπισκότο ριζιού έχει 15 γραμμάρια, ε, πάντα. Ε, έτσι κυκλοφορεί. Μια φρυγανιά ατομική είναι κάτω από 100 γραμμάρια. Όλα αυτά βέβαια είναι μια κάποια καινοτομία, συνάδελφοι. Πάντως είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν προταθεί μέχρι τώρα. Με την κυρία Σόμερς τα συζητάει η Αρμόδια Επιτροπή και στην ΙΜΚΟ επίσης, αλλά δεν αναφέρονται στις εκθέσεις τους. Το GTM επίσης, η μέση ποσότητα που συμβουλεύουμε στον καταναλωτή ημερησίως. Ναι, αλλά εξαρτάται ποιος Γιατί μπορεί μία να είναι έγκυος, μία άλλη να είναι πολύ ηλικιωμένη που να χρειάζεται περισσότερο ασβέστιο, μπορεί να είναι ένα παιδάκι τριών χρονών. Ε, δεν μπορούμε αυτό εύκολα να το πούμε. Αλλά δίνει ένα μέσο όρο, α πούμε. Αλκοολούχα ποτά τώρα. Εδώ νομίζω ότι έχουμε διαφορετική ρύθμιση. Οπότε το 1,2% ενόπνευμα πρέπει να το διατηρήσουμε. Μία εξαίρεση θα έκανα για τα αλκοπόψ που είναι μεικτά ποτά που περιέχουν ενόπνευμα που τα πουλάει βιομηχανία στους νέους σαν λεμονάδες, αλλά που έχουν. Ε, δεν είναι μόνο η βότκα, μπορεί να είναι μπακάρι. Α, συγγνώμη, δεν πρέπει να λέω εδώ πέρα. Μάρκες, εν πάση περιπτώσει. Είναι πάνω από το μέσο όρο της μπύρας, αλλά πουλούνται σαν αναψυκτικά. Για τους νέους, καλά δεν λέω ότι είναι εγκληματικό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι σωστό. Γιατί ξέρουμε ότι το πρόβλημα του αλκοόλ είναι μεγάλο μεταξύ των νέων. Αν ε, στις διαφημίσεις θέλουν να το περάσουν σαν ε, αναψυκτικό, ε, το Alcopops είναι ένα μεικτό ποτό, ακριβώς, που περιέχει και ενόπνευμα και αναψυκτικό. Δεν είναι βέβαια μέσα ούτε το κρασί, που έχει μυρουδιά κρασιού, δηλαδή ένα προϊόν μπύρας. Πάντως έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ενόπνευμα και δεν πρέπει να μείνουν έτσι. Τα μη προσυσκευασμένα τώρα τρόφιμα. Ε, εννοείται, αν πάτε στο χασάπι και του πούτε ε, να σας κόψει μια μπριζόλα, πώς θα σας πει τώρα ακριβώς πόσοι, πόσες ε, θερμίδες έχει. Ε, σίγουρα, αν δείτε ότι υπάρχει περισσότερο λίπος, εννοείται ότι και οι θερμίδες θα είναι παραπάνω. Και για τα εστιατόρια, Επίσης δεν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε σε αυτή τη ρύθμιση, τη μελλοντική ρύθμιση. Τέλος, δεν μιλάω γι' αυτό στην εκθεσή μου, γιατί ακριβώς είμαι κατά. Πρόκειται την απλοποίηση μέσω των διαφορετικών χρωμάτων, όπως στο φανάρι στην κυκλοφορία. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να απλοποιούμε την ενημέρωση, να την καταλαβαίνει καλύτερα χωρίς όμως να τον οδηγούμε σε λάθη. Γιατί άμα βάλουμε πως είναι τα φώτα της κυκλοφορίας, δηλαδή ότι είναι πιο ανοιχτόχρωμο, ε, δεν έχει ξέρω ή... Υπάρχουν όμως και τα προϊόντα, τα οποία και αυτά θα δημιουργήσουν ε, μπέρδεμα στον καταναλωτή. Γιατί υπάρχουν ε, πραγματικά προϊόντα που δεν είναι ερζάτς, τα οποία μπορεί να έχουν λίπος, αλλά είναι καλά. Ενώ με αυτό το σύστημα... Να, η Coca-Cola, η Light θα έχει πάντα πράσινο, ενώ το γάλα το πλήρες θα είναι πορτοκαλί ή κόκκινο. Ε, δεν νομίζω ότι θα ήταν σωστή μια τέτοια πληροφορία εντό εγωγικών προς τον καταναλωτή. Σίγουρα θα μας δοθεί ξανά η ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτά και να κάνουμε και τροπολογίες. Πάντως για τις τροπολογίες, τουλάχιστον 30 έχω συμπεριλάβει από την παλιά έκθεση. Δεν θέλω να αποφύγω τη συζήτηση, κάθε άλλο, αλλά από την άλλη μεριά θέλω να κατακλειστώ από τροπολογίε, γιατί δεν νομίζω ότι θα ήταν καλό, θα βοηθήσει στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μάρκ. Το θέμα είναι σημαντικό και υπάρχουν αρκετές τροπολογίες. Το περίμενα, θα έλεγα. Ας ξεκινήσει η συζήτηση, έχουν εγγραφεί αρκετοί. Γι' αυτό θα ήθελα να μην μακρηγορήσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ταραμπελά για μια εξαιρετική έκθεση και για τις πρωτοβουλίες που πήρε για τη διεύρυνση της εμβέλειας ακριβώς των προϊόντων τα οποία καλύπτει το θέμα της ονομασίας και χώρας προέλευσης έχει μεγάλη σημασία για τον καταναλωτή αλλά ιδιαίτερα για τον παραγωγό, ιδιαίτερα για τους καλούς παραγωγούς τους οποίους θα ευνοήσει η καταγραφή, η αναγραφή μάλλον της προέλευσης του προϊόντος. Έχω ένα ερώτημα γιατί ίσως δεν έχω διαβάσει προσεκτικά την πρόταση. <clears throat> Τι κατάσταση έχει δημιουργηθεί σχετικά με τα μη γενετικά τροποποιημένα προϊόντα ρυθμίζεται, ορίζεται. Ένα άλλο θέμα αφορά τις ετικέτες για προϊόντα τα οποία βασίζονται στην ζωική παραγωγή σχετικά με τον τρόπο σφαγής. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο ήμουν εισηγητής για την σφαγή των ζώων και είχαμε συζητήσει τα διάφορα, τις διάφορες μεθόδους φαγής ε, που ακολουθούνται. Ξέρετε τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν για θρησκευτικούς λόγους. Αυτά τα θέματα τα έχει λάβει υπόψη του κύριο Σταραμπελά. Ευχαριστώ. Paulsen. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή, διότι νομίζω ότι οι προθέσεις που έχει περιλάβει στην έκθεσή του και οι ιδέες του είναι ορθές. Συμφωνώ με αυτό το σύστημα του σηματοδότη, που, με αυτά που είπατε για το σύστημα του σηματοδότη. Θεωρώ ότι είναι ανοησία, σαν χλαμάρα. Όλη αυτή η ιστορία με τα 100 γραμμάρια ή τα 100 χιλιοστά του λίτρου είναι ένα απλό σύστημα και δεν νομίζω ότι οι πολίτες στην Ευρώπη είναι τόσο ανόητοι ώστε να μην μπορούν να κάνουν την πρόσθεση ή την διαίρεση με εκατοστίες μονάδες. Και αν μιλούμε επιτέλους για εμπιστοσύνη των καταναλωτών, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να κάνουμε. Εάν έχετε έναν εύρωστο άνθρωπο ο οποίος ζυγίζει 100 κιλά, χρειάζεται 2.800 θερμίδες την ημέρα, να καταναλώνει δηλαδή, για να διατηρήσει το βάρος του και τη ζωή του. Εάν έχετε έναν άνθρωπο 70 κιλών θα δείτε αναλογικά ότι έχει ανάγκη από 1950 θερμίδες. Αν μιλούμε για έναν ευρωβουλευτή θα δείτε ότι δεν χρειάζεται τόσες πολλές θερμίδες για να κάνει την δουλειά του. Αν είσαι όμως ξυλοκόπος ή κάτι παρόμοιο, χρειάζεστε βέβαια πολύ περισσότερες θερμίδες για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες του επαγγέλματος και για να μπορέσετε να επιβιώσετε δηλαδή. Νομίζω λοιπόν ότι έχει μεγάλη σημασία να είμαστε αυστηροί και να τηρήσουμε αυστηρά ένα απλό σύστημα υπολογισμού του, της περιεκτικότητας σε θερμίδες των διαφόρων τροφίμων. Σας ευχαριστώ κυρία Πάουλσεν. Η κυρία Ρέιμερς. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ταραμπέλα για την έκθεσή του. Δεύτερον, θέλω να τονίσω ότι είναι καθήκον μας να φροντίσουμε ώστε ο, να ο καταναλωτής να διαθέτει υπαρκείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο τρόφιμο. Παρ' όλα αυτά, οι διάφορες επισημάνσεις με ετικέτες κλπ. δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν υπερβολικά τον παραγωγό και την βιομηχανία. Γι' αυτό θεωρώ ότι ορισμένες προσεγγίσεις της εκθέσεως είναι αξιοπρόσεκτες και πρέπει να υποστηριχθούν, άλλες θεωρώ ότι είναι υπερβολικές. Σωστό βρίσκω να αναγράφονται οι περιεκτικότητες ανά 100 γραμμάρια ή ανά 100 ε, χιλιοστά του λίτρου. Σημαντικό είναι επίσης για μη τυποποιημένα προϊόντα να εξαιρεθούν από τον κανονισμό. Πάλι για μη τυποποιημένα προϊόντα θα πρέπει να διατίθεται οι πληροφορίες στον καταναλωτή ε, σχετικά με την προέλευση του προέδρου κτλ. εφόσον αυτός θέσει την ερώτηση. Συμφωνώ λίγο πολύ με, τα, με την κριτική για το σύστημα του σηματοδότη. Είμαι και κατά των ε, ιδιαιτέρων εθνικών κανόνων για θέματα επισήμανσης με ετικέτες. Ε, θεωρώ επίσης ότι είναι σωστό να γίνει εκπαίδευση των καταναλωτών, να ληφθούν δηλαδή ιδιαίτερα μέτρα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν σωστά τις διαθέσιμες πληροφορίε οι καταναλωτές. Νομίζω ότι ο κ. Ταραβέλα έχει συντάξει καλά το σχέδιο, έχει βάλει σωστά ιδίω στο επίκεντρο του ενδιαφέροντο τα αγροτικά, αλλά υπάρχουν και ορισμένε παγίδε για την αγροτική παραγωγή. Για παράδειγμα, η ένδειξη προέλευσης δεν μπορώ να δεχθώ υποχρεωτική ένδειξη, διότι αυτό οδηγεί ξεκάθαρα σε ένα μειονέκτημα για τον παραγωγό. Διότι αφαιρείται από τον παραγωγό ένα, ένα εργαλείο του marketing. Διότι εφόσον είναι επιθυμητή η ένδειξη της ε, προέλευσης, έχει τη δυνατότητα να έχει ένα πλεονέκτημα για τη διάθεση στην αγορά ο καταναλωτής. Εγώ λοιπόν προτιμώ να υπάρξει εθελοντική ε, ένδειξη της προέλευσης. Στην περίπτωση υποχρεωτικής ένδειξης προέλευσης υπάρχει και το πρόβλημα της εφαρμοσιμότητας. Υπάρχουν σήμερα τροφήματα, δε, συγγνώμη, τρόφιμα τα οποία συναπαρτίζονται από πολλά μέρη και αυτά αλλάζουν. Καμιά φορά η προμήθεια του καταστήματος γίνεται από μια, ή του, ή ε, μεταποιητή γίνεται από μια περιφέρεια, άλλη φορά γίνεται από άλλη, αλλάζουν ε, τα συστατικά και όλα αυτά σημαίνουν βέβαια τεράστια επιβάρυνση για τους μεταποιητές. Ένα άλλο πρόβλημα που έχω είναι το κοινοτικό σύμβολο της ε, πλεονεκτικής διατροφής. Βρίσκω πρόβλημα να υπάρχει εδώ όπως και το σύστημα του σηματοδότη. Θεωρώ ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι ο ίδιος σε θέση να κρίνει ποια τρόφιμα θέλει να προμηθευτεί και να καταναλώσει. Δεν θέλω να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καθήκον να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ως ή τα τρόφιμα ως καλά ή όχι για την υγεία του καταναλωτή. Προτιμώ ο καταναλωτής να τα αξιολογεί μόνος του. Τώρα, για το, μέθοδο, για το μέγεθος των στοιχείων, των γραμμάτων και ψηφίων, θα προτιμούσα να ξεκαθαρίσουμε ότι πρέπει να υπάρχει αντίθεση και των χρωμάτων μεταξύ γραμμάτων και φόντου. Εάν πρέπει εάν δεχθούμε ανά 140 ε, τετραγωνικά εκατοστά 22 χιλιοστά ε, γράμματα εκεί βρίσκω ότι υπάρχει πρόβλημα γιατί θα είναι πάρα πολύ πυκνά τα γράμματα. Τώρα, για τα αναψυκτικά που περιέχουν και ενόπνευμα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπουν εδώ. Μπορούμε να ενημερώσουμε την νεολαία πολύ καλύτερα με ειδικά προγράμματα και όχι να δηλώσουμε πάνω στις συσκευασίε των αλκοπόψ. Άλλωστε από την δική μου εμπειρία ως νεαρά, από νεαρά ηλικία δηλαδή, και από τις αναστροφές με τους φίλους μου διαπίστωσα ότι όλοι εν τέλει προτιμούσαν τα αναπτυκτικά που είχαν υψηλότερο περιεχόμενο σε ενόπνευμα και αυτά έπαιρναν από τα ράφια των καταστημάτων. Πρέπει να σκεφτεί κανείς και ως νέος στην περίπτωση αυτή και ότι θέλουν να εντυπωσιάσουν τους συνομιλίκους τους. Ευχαριστώ. Ο Αλβέρτος Ντες. Χωρίς μικρόφωνο κύριο Ντες. Συγγνώμη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Ταραμπέλα για την υποβολή της εκθέσεως και για τις λογικές ε, προτάσεις που έχει κάνει. Πρόσφατα μας και προσκαλέσει στην περιφέρειά του, όπου μεταβήκαμε μαζί με άλλα μέλη της ε, Επιτροπής και θαυμάσια προϊόντα μπορέσαμε να γευθούμε εκεί επί τόπου. Μου άρεσε ότι είναι αντίθετος με το σύστημα του σηματοδότη. Είναι πραγματικά τεράστια ανοησία. Φανταστείτε να πηγαίνετε να, να κινείστε προς την κατεύθυνση μια μεγάλη διασταυρώσεως και να βλέπετε εκεί πέντε ή έξι σηματοδότες οι οποίοι να δείχνουν όλοι διαφορετικά πράγματα. Το ίδιο θα συμβεί και με την επισήμανση των τροφίμων. Εγώ θέλω να υπάρχουν λογικές πληροφορίες, αλλά όχι όμως τέτοια παραπλάνηση. Θυμίζω και το παράδειγμα του Έλμαρ Μπροκ, που σίγουρα ζυγίζει παραπάνω από 100 κιλά και είπε αυτός ότι του αρέσει το σύστημα του σηματοδότη γιατί τότε θα πάρει αμέσως τα προϊόντα που έχουν απάνω το κόκκινο, διότι αυτά προτιμάει. Ε, θέλω επίσης να πω και κάτι πιο σοβαρό τώρα. Η μητέρα μου που μόλις έκλεισε τα 86 χρόνια ηλικίας με παρακάλεσε να πάω να επισκεφθώ μία θεία μου 94 ετών αυτή στο Μόναχο. Δεν την έχω δει ποτέ στη ζωή μου τη γυναίκα αυτή. Πήγα λοιπόν να την επισκεφθώ, χτύπησα το κουδούνι, εμφανίζεται μία κυρία που λέω αποκλείεται να είναι του τυδό διότι αυτή είναι το πολύ 70. Ήταν όμως η θεία μου 94 ετών και μου είπε έλα να διπνήσουμε μαζί. Λίγο πριν είχα δει στην βαβαρική τηλεόραση μία ε, γιατρό που εξηγούσε πόσο κακό είναι να τρώει κανείς λιπαρό κρέας, ότι είναι περίπου αυτοκτονία. Αυτή λοιπόν η θεία μου, μεγάλη θεία δηλαδή, με προσκάλεσε να καθίσω να γευθώ μαζί της το κρέας και βλέπω να αφαιρεί το λίπος και λέω θα είδε και αυτή την ίδια εκπομπή. Όμως αυτό που έκανε ήταν να αφαιρέσει το στεγνό κρέα και να κρατήσει το λίπο. Και μου είπε ότι ποτέ στη ζωή τη δεν έχει φάει το στεγνό κρέα, το οποίο βρίσκει άγευστο. Σκέφτηκα λοιπόν και εγώ, θα έπρεπε να ήταν εδώ η γιατρό τη ε, τηλεοράσεω εχθέ, διότι αμέσω θα πάθαινε ε, καρδιακή προσβολή όταν την έβλεπε να κάνει τέτοια πράγματα. Θαυμάσια, Άλμπερτ. Η κυρία Ελάνη Γκαρσία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον κύριο Ντές για το ωραίο αυτό που μας είπε. Τώρα, στην ε, έκθεση αντικτύπου που ακόμα δεν έχουμε, θα ήταν πολύ σημαντικό να την είχαμε γιατί μερικές φορές βάζουμε στις ετικέτες πράγματα που δεν είμαστε σίγουροι ότι τα καταλαβαίνουν ή τα θέλουν οι καταναλωτές. Τώρα για τον κύριο Ταραβέλα, τι έχω να πω. Ένα κύριος πράγμα. Όταν μιλάμε για την προέλευση των προϊόντων, υπερβάλλουμε με τις απαιτήσει μας. Τι εννοώ. Ας υποθέσουμε, έχουμε λοιπόν κάποιον που παράγει είναι φρυγανιές και ξηρούς καρπούς. Αν λοιπόν πούμε ότι πρέπει να ξέρουμε κάθε ένας από τους ξηρούς καρπούς από πού προέρχεται, που βάζει μέσα στα μπισκοτάκια του ας πούμε, ε, πώς θα το κάνουμε αυτό. Γιατί αν κάποιος πρέπει κάθε φορά που αγοράζει ε, καρύδια, αμύγδαλα, δεν ξέρω εγώ τι, να αλλάζει και την ετικέτα στο προϊόν του, ε, καήκαμε. Λοιπόν, το να λέμε ότι είναι κοινοτική προέλευση, αυτό φτάνει. Γιατί έτσι ενισχύεται και η ιδέα τη ενιαία αγορά. Μην το ξεχνάμε. Και είναι στην πράξη πολύ πιο αποτελεσματικό. Και επιπλέον, το να ξέρει κανεί ότι είναι κοινοτική προέλευση, ε, βοηθάει και στην εικόνα τη Ευρώπη. Αλλιώ είναι σαν να λέμε στον ε, παραγωγό κάθε φορά που βάζετε ξηρού καρπούς στα μπισκότα σα πρέπει να τα από το ίδιο μέρο για να κρατάτε την ίδια ετικέτα και να μην την αλλάζετε κάθε τρει και λίγο. Τώρα στη συνάδελφο όταν πάει σε, στο σούπερ μάρκετ ένας νέος και δει ότι κάπου έχει περισσότερο αλκοόλ, όντως φέρτο, φέρτο θα λέει. Αλλά αν το κάνουμε αυτό με τα αλκοπόψ, πρέπει να το κάνουμε με όλα. Γιατί δεν υπάρχουν και λικέρ κάποιων προϊόντων που να έχουν ε, τουλάχιστον τόση ζάχαρη και τόσο αλκοόλ όπως και τα αλκοπόψ. Οπότε τα αλκοπόψ είναι ένα επιπλέον αλκοόλ. Σωστά τα έχουμε βγάλει. Γιατί δεν πρέπει εδώ να τα εξετάζουμε σε αυτή την έκθεση. Αλλά εγώ θα έβγαζα και κάθε μνήα ε, σε αντίστοιχα προϊόντα στην οδηγία αυτή και στον κύριο Βασικόφσκι που αναφέρθηκε στα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Αν έχουμε τέτοια απέτηση από τρίτες χώρες, καλώς. Αν όμως δεν την έχουμε, να μην την έχουμε ούτε από τους κοινοτικού ε, παραγωγούς. Δεν μπορεί να βάζουμε τέτοιες υποχρεώσεις στους κοινοτικού παραγωγούς που δεν τις βάζουμε στους άλλους. Ο κύριος Γιάρα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον κύριο Ταραμπέλα για την έκθεσή του. Νομίζω ότι διαγράφεται μια τάση στην ε, Επιτροπή Γεωργίας, ναι μεν για την επισήμανση, θα δούμε βέβαια τι ακριβώς σημαίνει, αλλά πάντως τα χαρακτηριστικά να είναι επαρκείς πληροφορίες αλλά όχι γραφειοκρατία. Οι καταναλωτές άλλωστε έχουν ε, διαφορετικές ανάγκες ενημέρωσης. Υπάρχουν καταναλωτές οι οποίοι θέλουν να γνωρίζουν τα πάντα, Υπάρχουν άλλοι που απλώ του ενδιαφέρει εάν είναι γευστικό το προϊόν ή όχι. Εγώ, ε, για παράδειγμα, δεν ε, ε, έχω τόσο μεγάλη ανάγκη να έχω όλες τις λεπτομέρειες. Γι' αυτό προτιμώ να είναι γευστικά τα προϊόντα. Πρέπει βέβαια να φροντίσουμε ανεξαρτήτως του τι θα βάλουμε στην ετικέτα και πώς θα γίνει δηλαδή γι' αυτό με πόσες λεπτομέρειες κτλ. Χρειαζόμαστε ενημέρωση διατροφής. Άλλωστε υπάρχει και επιστήμη της διατροφής. Χρειαζόμαστε ενημέρωση διατροφής για τους νεαρούς και τις νεαρές μας να γνωρίζουν τι σημαίνει η υγιεινή διατροφή. Να φροντίσουν να το συνδυάσουν και με επαρκή άσκηση διότι όσο περισσότερο καταναλώνω τόσο περισσότερο πρέπει να κινούμε. Και σε ό,τι αφορά το σύστημα του σηματοδότη, ναι μεν είναι ελκυστικό από πρώτη άποψη, αλλά στην πραγματικότητα είναι ανόητο. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε και άλλη ενημέρωση, πρέπει να περάσει και μέσα από τη σχολική εκπαίδευση. Δεν λύνονται τα προβλήματα μοναχά με την ετικετοθεσία. Πάρτε το παράδειγμα των σιγαρέτων. Το γράψαμε απάνω και με μεγάλα στοιχεία ότι είναι επικίνδυνο. Όσοι καπνίζουν εξακολουθούν να καπνίζουν. Ενημέρωση χρειάζεται, εκπαίδευση χρειάζεται. Αυτό ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά. Χόισλινγκ. Συμμερίζομαι τα πολυάριθμα συγχαρητήρια προς τον κύριο Ταραμπέλα και εμένα μου αρέσει η εκθεσή του. Από την αγροτική σκοπιά θέλω να τονίσω ορισμένα πράγματα ακόμα. Είμαι υποχρεωμένο να αντίπω στην συνάδελφο μου Ράιμερ, αν και δεν μου αρέσει. Εγώ θεωρώ ότι είναι, πρέπει να είναι υποχρεωτική η ένδειξη προέλευση. Μόνο τότε έχει κάποιο νόημα. Διότι εφόσον θέλουμε να διατηρήσουμε μια περιφερικότητα, εφόσον θέλουμε να διατηρήσουμε ένα, να επιτύχουμε ένα περιορισμό των διοξιδίων του άνθρακα, Πρέπει να τονίσουμε την περιφερικότητα, πρέπει να τονίσουμε την προέλευση από κάποια συγκεκριμένη περιφέρεια και πρέπει αυτό να το καταλαβαίνει ο καταναλωτή. Το ίδιο πρέπει να ε, ε, επιβληθεί και στα προϊόντα κρέατο, κρέα και προϊόντα κρέατο. Διότι εκεί που βρισκόμαστε τώρα, το μόνο που ενδιαφέρει είναι το προϊόν να είναι φθηνό, ανεξαρτήτως του πόσο μακριά ταξιδεύει. Δεύτερο, η δυνατότητα μη τυποποιημένων προϊόντων να χαρακτηρίζονται επιτόπου. Είναι δυνατόν σε καταστήματα να γίνεται με καταλόγους, με λίστες. Αυτό είναι δυνατόν. Υπάρχουν και παραδείγματα. Και δεν νομίζω ότι αποτελεί ιδιαίτερη επιβάρυνση για τον ε, μεταποιητή ή τον έμπορο. Τώρα, για, την, για τους μικρούς παραγωγούς. Ασφαλώς δεν πρέπει να επιβαρυνθούν με πρόσθετη γραφειοκρατία. Αυτό μπορεί να γίνει εφόσον διαθέτουν τα προϊόντα τους σε περιφερειακές αγορές. Και μια ακόμη πρόταση. Έχουμε επισήμανση στα αυγά. Και έχουμε επιτύχει, έχουμε καταφέρει μεγάλες επιτυχίες για τα αυγά που καταναλώνουν ε, οι, άνθρωποι στο πρωινό τους. Έχουμε δει να στρέφονται σε κατανάλωση αυγών που δεν προέρχονται από συστοιχίες κλωβών ορνήθων. Θα πρέπει το ίδιο να γίνει και στα προϊόντα όπου βρίσκονται μέσα αυγά. Δεν είναι μόνο δηλαδή καθαρά τα αυγά, αλλά σε προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τους αυγά. Θα πρέπει και εκεί να μπει ο χαρακτηρισμός του αυγού ως προερχόμενο από ε, όρνηθες ελεύθερας βοσκής. Ελευθερας βοσκής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Να κάνω δύο παρατηρήσεις. Δεν ξέρω πόσοι από εμά στην αίθουσα βλέπουν τακτικά τις ετικέτες όταν πηγαίνουν να αγοράσουν ε, κάποια προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Εγώ μέχρι πριν 15 μέρες τρεις εβδομάδες άντε, όταν άρχισα να παίρνω κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες, δεν το έκανα. Εδώ και λίγες μέρες προσπαθώ να διαβάζω τις ετικέτες, είναι περίπλοκο, δυσανάγνωστες και γενικά οι πληροφορίες τις οποίες περιέχουν δεν είναι, ε, θα έλεγα, αφομοιώσιμες από τον καταναλωτή παρατήρησα στο κατάστημα για να δω πόσοι από αυτούς που αγόραζαν διάβαζαν τις ετικέτες. Πολύ λίγοι. Τι θέλουμε λοιπόν. Θέλουμε να ηθικοποιήσουμε θα έλεγα την αγορά. Να γνωρίζουμε τι υπάρχει μέσα στο πακέτο. Αυτός ο στόχος είναι διαφορετικός από τον στόχο της υγείας και της εκπαίδευσης του καταναλωτή. Για 13 χρόνια ήμουν δημοτικός σύμβουλος σε μια μεσαία γαλλική πόλη με πολλά κοινωνικά προβλήματα. Το θέμα της κακής διατροφής και της έλλειψης διατροφικής ισορροπίας είναι κάτι το οποίο με απασχόλησε πολύ σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Τι κάναμε το σημαντικό. Συγκεντρώσαμε νοικοκυρές από οικογένειες αποσαφρωμένες θα έλεγα, των οποίων τα παιδιά παρουσίαζαν δείγματα κακής διατροφής και τους μάθαμε να μαγειρεύουν ισορροπημένα προϊόντα με, απλά, με απλές πρότεσίλες και διαπιστώσαμε έτσι πάρα πολύ σύντομα τα συγκεκριμένα παιδιά πήγαν καλύτερα ήταν πιο προσεκτικά και συγκεντρωμένα κτλ. Αν θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε την υγεία του καταναλωτή, θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναπτύξουμε συγκεκριμένες παιδαγωγικές δράσεις, όπως ας πούμε η διανομή φρούτων στα σχολεία κτλ. Αλλά να μην ανακατεύουμε τα πάντα, να μην μας λέγουν ε, σώνει και καλά ότι πρέπει να ελαφρύνουμε την ετικέτα για να ελαφρύνουμε τη συσκευασία, μειώνοντας ε, έτσι την ενημέρωση του καταναλωτή. Αυτή η κωδική με τις γραμμούλες που υπάρχουν στα προϊόντα θα πρέπει να μας λένε τα πάντα για το προϊόν. Το πότε έχει γίνει η παραγωγή του, που έχει γίνει η παραγωγή, τα συστατικά του. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προσφέρεται θα έλεγα δεν δημιουργεί προβλήματα και αυτοί οι οποίοι επιθυμούν να έχουν τις ετικέτες θα τις έχουν και στο σπίτι τους και στα καταστήματα όπως το επιθυμούν και όποτε το επιθυμούν. Δεν θα πρέπει να αναμίξουμε τους δύο στόχους γιατί αν το κάνουμε δεν θα ικανοποιήσουμε ούτε τους μεν ούτε τους δε. Ευχαριστώ Μίσελ Τόφμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα αυτά που είπε ο προηγούμενος ομιλητής και θα σταθώ λίγο σε αυτά. Συμφωνώ μαζί του. Εάν πράγματι ένας καταναλωτής μπει σε ένα υπερκατάστημα να κάνει τα εβδομαδιαία ψώνια, θα έλεγα, πρέπει να έχει ένα κάποιο επίπεδο ενημέρωσης. Δεν το έχει πάντα. Καμιά φορά είναι καλύτερα οι επισημάνσεις να έχουν λιγότερα παρά περισσότερα. Πρέπει να γίνει και μια διάκριση μεταξύ δυνητικών και υποχρεωτικών στοιχείων στην ετικέτα. Εάν οι παραγωγοί θεωρούν ότι είναι χρήσιμο και για τη διάθεση του προϊόντος του στην αγορά να μπουν κάποια πρόσθετα στοιχεία, αυτό να επιτρέπεται και να ελέγχεται βέβαια. Για παράδειγμα, ε, επισήμανση της προέλευσης του προϊόντος εάν έχει γενετικά τροποποιημένα, τροποποιημένους οργανισμούς στο περιεχόμενο του. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν ένα περιορισμένο αριθμό καταναλωτών. Και επισημαίνω ότι εάν τα πάρουμε πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα σημαίνουν και αύξηση της γραφειοκρατίας γιατί πρέπει και να ελέγχονται. Πρέπει να υπάρξουν δηλαδή και συστήματα ελέγχου. Δεν μπορεί απλώς ο κάθε παραγωγός να γράφει επάνω στο προϊόν ό,τι θέλει. Τώρα κάτι που είπε και ο κύριο Χόισλινγκ προηγουμένω, Για μικρούς παραγωγούς να υπάρξουν εξαιρεσει. Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι επιθυμούμε να ενισχύσουμε την άμεση διοχέτευση ε, στις αγορές, την άμεση διάθεση στις αγορές. Εάν θέλουμε να του φορτώσουμε και άλλες τέτοιε επιβαρύνσεις, τότε του ε, κόβουμε κυριολεκτικά τα πόδια. Πρέπει να υπάρξουν λοιπόν κάποιε αποκλήσεις υπέρ αυτών. Κάτι που είπε η κυρία Ράιμερ προηγουμένω σε σχέση με τον σηματοδότη. Η έκθεση προβλέπει την εισαγωγή μιας ετικέτας για ιδιαίτερα υγιεινά προϊόντα. Αυτό είναι να ανοίγουμε ένα παραθυράκι πάλι στο σηματοδότη. Ήδη ο Παράκελσος προαιώνων είχε πει ότι αυτό που σε, μικρή, σε μεγάλη δόση είναι δηλητήριο, σε μικρή δόση μπορεί να είναι φάρμακο. Ένα ποτηράκι κρασί σας κάνει καλό. Αν πιείτε τρία μπουκάλια κρασί, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Το να πει κανείς τώρα τούτο το τρόφιμο είναι υγιεινό, τούτο δεν είναι κτλ. Αυτά είναι ανοησίες, ούτε εξυπηρετούν τον καταναλωτή και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να το αποτρέψουμε, να το αποκλείσουμε σωστά αυτά που λέτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να εκπαιδεύσουμε σωστά μέσω των ετικετών τους καταναλωτές. Δεν θα δουλέψει αυτό, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οι ετικέτες μπορούν να βοηθήσουν λίγο, αλλά δεν μπορούν σίγουρα να υποκαταστήσουν τις δημόσιες πολιτικές για την ενημέρωση και την παιδεία. Να διευκρινίσουμε επίσης ότι, και η, ότι η ιδέα των σηματοδοτών είναι εντελώς απαράδεκτη. Για την παρουσίαση την ποσοτική των συστατικών αυτό είναι κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Η βιομηχανία έχει εν μέρει ανταποκριθεί σε σχέση με αυτά τα οποία ζητάμε. Αναφέρθηκε η κυρία Χεράντζ Γκαρσία στο ότι η έρευνα στο τι θέλουν οι καταναλωτές τις ετικέτες δεν έχει ολοκληρωθεί. Και εμείς εδώ αποφασίζουμε το τι θα μπει στις ετικέτες χωρίς να είμαστε ενήμεροι. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό να κάνουμε αυτό το οποίο προσπαθούμε. Το δεύτερο σημείο για τις ονομασίες προέλευσης. Εκεί που υπάρχει θέμα είναι ότι πολλές φορές οι καταναλωτές λέγουν ας πούμε Ιρλανδικός καπνιστός Σολομός ή καπνιστός Ιρλανδικός Σολομός. Ο ένας είναι Ιρλανδικός, ο άλλος δεν είναι. Όλοι υποθέτουν όμως ότι και στις δύο περιπτώσεις είναι Ιρλανδικός. Οι ετικέτες δηλαδή πολλές φορές είναι παραπλανητικές. Νομίζω ότι μπορούμε να φανούμε πιο λιγότερο φιλόδοξοι και πιο συγκεκριμένοι σε σχέση με το τι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ο Λένις Ιακ. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτούς οι οποίοι ε, συνεχάρισαν τον εισηγητή και να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, οι ετικέτες σχετικά με την προέλευση των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τα μεταποιημένα. Οι πρώτες ύλες δηλαδή. Καλό θα ήταν, σαν παράδειγμα στις Μαρμελάδες, στην Πολωνία, στην Ιταλία, στις άλλες χώρες, να μπορούμε να δούμε πράγματι από πού προέρχονται οι φράουλες. Είναι ευρωπαϊκές φράουλες ή μήπως οι φράουλες αυτές είναι φράουλες εισαγωγής, αλλοδαπές. Ο καταναλωτής πρέπει να μπορεί να αποφασίσει αν επιθυμεί τις κινέζικες φάουλες ή τις ευρωπαϊκές φάουλες. Όταν μιλάμε για συνειδητή καταναλωτική και αγοραστική συμπεριφορά, θα πρέπει να γνωρίζουμε. Αν ας πούμε εγώ παραγγείλω κάπου μύδια, πρέπει να γνωρίζω αν είναι ευρωπαϊκά μύδια ή αν είναι εισαγόμενα μύδια από μακρινές περιοχές του κόσμου. Αυτές είναι οι πληροφορίες οι οποίες θα βοηθήσουν έτσι ώστε να κάνω μια σωστή ενημερωμένη επιλογή. Να πω επίσης ότι οι πληροφορίες αυτές, αυτού του είδους οι πληροφορίες, έχουν μεγάλη σημασία για συνειδητοποιημένους καταναλωτές που έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν όταν έχουν χρήματα βέβαια. Και εδώ ακούγονται κάποιες φωνές που λέγουν ότι στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί συμπολίτε μας οι οποίοι στα καταστήματα δεν κοιτούν παρά μόνον την τιμή και δεν ασχολούνται με αυτά τα οποία εμείς συζητάμε σήμερα όταν αγοράζουν κάτι. Δεν κοιτούν αν είναι υπερθερμιδικό ή αν έχει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες ζάχαρης. Πολλές φορές η πλειοψηφία θα έλεγε κανείς των Ευρωπαίων ασχολούνται με το ότι ίσως κάποια προϊόντα να μην είναι τόσο πλούσια σε ζάχαρη, θερμίδες και βιταμίνες πριν τα αγοράσουν. Οι πληροφορίες λοιπόν, οι οποίες αυτή τη στιγμή πρέπει να περιλαμβάνονται στις ετικέτες, είναι σημαντικές για να είναι ενήμερος ο αγοραστής αυτών που έχουν χρήματα. Αυτοί οι αγοραστές που έχουν χρήματα βέβαια και έχουν την δυνατότητα να κάνουν τις επιλογές. Το θέμα είναι τι θα μπορέσουμε να κάνουμε έτσι ώστε οι ετικέτες και τα προϊόντα να περιλαμβάνουν ξεκάθαρα στοιχεία τα οποία να αφορούν και αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες αγοράς και σωστής επιλογής. Και τι μπορούμε να κάνουμε για τον καταναλωτή όταν έχει μπροστά του δύο ταυτόσιμα προϊόντα και δεν κοιτά μόνο την τιμή, κάτι το οποίο είναι 2% φτηνότερο ή 5% ακριβότερο, αλλά μέσω των πληροφοριών στις ετικέτες να επιλέγει το προϊόν το οποίο ίσως να είναι ο λίγο ακριβότερο αλλά είναι ευρωπαϊκό προϊόν και με καλύτερη διατροφική αξία. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος τον οποίο θα επιλέξουμε. Ευχαριστώ. Ας κλείσουμε λοιπόν τον κατάλογο των ομιλητών. Άγνα. Ας πούμε ότι είμαι η κυρία Σμιθ που τη στήθηκε να φτιάξει ένα γλυκό για ένα φιλανθρωπικό χώρο. Η κυρία Σμιθ φτιάχνει καλά κέικ. Το πρόβλημα στο κέικ είναι ότι δεν υπάρχει ένα κυρίαρχο συστατικό. Βάζει λοιπόν αλεύρι. Θα μιλήσει τώρα για τους κινδύνους του γλουτενίου. Βάζει και αυγά. Τα αυγά είναι από όρνηθες ελεύθερης βοσκής. Έχουν φάει καλαμπόκι γενετικά τροποποιημένο, βάζει και μερικά καρύδια, προκαλούν αλλεργίες τα καρύδια. Βάζει και κεράσια. Είναι εισαγωγή από πού έχουν ε, προέλθει. Βάζει και ζάχαρη. Από πού προέρχεται, από ζαχαροκάλαμο ή από τέφτλο. Εάν καθίσει να τα σκεφτεί όλα αυτά τα πράγματα, το κέικ τελικά δεν θα γίνει και όλοι θα χάσουν γιατί θα ήταν και το πιο νόστιμο. Α δούμε λοιπόν τα πράγματα αυτά στο πιο βασικό επίπεδο και α μην τρομάζουμε και αποτρέπουμε τον κόσμο από το να κάθεται να φτιάξει ωραία και νόστιμα πράγματα. Δεν θα πρέπει να δημιουργούμε... Δεν θα πρέπει να δημιουργούμε περαιτέρω συγχύσεις στην προσπάθειά μας να δώσουμε τις σωστές πληροφορίες. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της, στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αναπληρώτηρα Γενική Διευθύντρια. Θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες πρώτες απαντήσεις. Θεωρούμε ενδιαφέρουσα την έκθεση του κ. Ταραμπέλα. Εν πωλής υποστηρίζει τις προτάσεις μας ιδιαίτερα στους τομείς τους οποίους θεωρούμε ότι είναι σημαντικοί. Το ότι υπάρχει διατροφική ε, ετικετοθεσία στην πρόσωψη σε εισαγωγικά στην εμπρόστια πλευρά της συσκευασία είναι κάτι το οποίο ήδη θεωρητικά έχει γίνει υποχρεωτικό και είναι κάτι επίσης το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την εκπαίδευση του καταναλωτή, η οποία πρέπει να συνεχίζεται παράλληλα έτσι ώστε ο καταναλωτής που είναι σε θέση και μπορεί να το κάνει να κάνει τις σωστές επιλογές προς την ευχαρίστησή του και για να προστατεύσει την υγεία του. Γι' αυτό αυτά τα οποία είπατε επίσης για τα αλλεργογόνα έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όπως επίσης και για το ότι ακόμα και αν ο εισηγητής δεν δέχεται την υποχρέωσή μας για τα 3 μιλιμέτρα, είναι σαφές ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα των ετικετών, γιατί πάρα πολλές φορές σχολιάζεται ότι οι ετικέτες είναι δυσανάγνωστες. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και την αντίθεση των χρωμάτων και το μέγεθος των γραμματοσυρών. Και έτσι θα μπορέσουμε ε, μέσω των προσπαθειών που κάνουμε να καταλήξουμε σε ένα καλό συμβιβασμό για την ετικετοθεσία των αλκοολούχων. Όλα τα αλκοολούχα προϊόντα εκτός από το κρασί, την πύρα και τα υνοπνευματόδη υποβάλλονται ε, στην υποχρεωτική ετικετοθεσία των συστατικών. ένα χυμός φρούτων, σαν παράδειγμα, πρέπει να λέει από τι αποτελείται και τη διατροφική του αξία. Αν προσθέσω λίγο υνοπνεύμα σε αυτή την περίπτωση εξαιρείται ένα τέτοιο προϊόν από την υποχρέωση ε, αναγραφής. Τώρα θα πρέπει να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις έτσι ώστε να υφίστανται όλα τα συγκρίσιμα προϊόντα αντίστοιχες υποχρεώσεις σχετικά με την αναγραφή επαναλαμβάνω των συστατικών. Σημειώσαμε τα σχόλιά σας για την προέλευση. Είναι σαφές ότι υπάρχει επιθυμία να καταγράφονται τα προϊόντα αυτά, ιδιαίτερα τα πρωτογενή προϊόντα. Εμείς σε σχέση με την πρόταση αυτή δεν έχουμε αλλάξει την άποψή μα ότι το καθεστώς αυτό παραμένει εθελοντικό, αλλά το έχουμε πλαισιώσει καλύτερα το καθεστώς αυτό, έτσι ώστε να δίδονται οι σωστέ πληροφορίες. Αλλά γύρω από αυτό το θέμα της προέλευσης, οι συνάδελφοι της ε, Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και η κυρία Φίσερ Μπόλ προσπαθούν να δουν ποια είναι τα βασικά γεωργικά προϊόντα στα οποία τεκμηριώνεται αν θέλετε η ανάγκη να υπάρχουν ετικέτες που να δηλώνουν την προέλευση για τις ημερίδες και την ημερήσια ποσότητα. Προφανώς είναι πολύ εύκολο να πει κανείς, αποφασίζουμε εξ αρχής ότι θα πούμε 5 μιλιλίτρι, 5 μιλιγράμμ. Αλλά μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε εναρμονισμένες μερίδες και όταν αυτό το κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τότε θα βελτιωθεί και η κατανόηση του καταναλωτή για τη σηματοδότηση Κατανάω ότι δεν συμφωνείτε εν πολύ. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πάρα πολλά σχήματα τα οποία αναπτύσσονται σε εθνικό επίπεδο και οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να βλέπουν να νιώθουν μια κάποια σύγχυση. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τον καταναλωτή και να επιδιώξουμε μια σταδιακή εναρμόνιση. Δεν λέμε τι πρέπει να κάνουμε από τώρα αλλά να δούμε τι ακριβώς είναι διαθέσιμο στην αγορά και να δούμε αν τα εθνικά σχήματα ενημέρωσης μπορούμε σταδιακά να τα εναρμονίσουμε. Θα ήθελα επίσης να διαβεβαιώσω τον τελευταίο ή τους τελευταίους ε, ομιλητές για να σας πω ότι η κυρία Σμιτ εξαιρείται της πρότασης. Μην ανησυχείτε όλες οι άμεσες τοπικές πωλήσει προϊόντων εξαιρούνται οι φιλανθρωπικές αυτές ε, οργανώσεις λοιπά Και συνεχώς η κυρία Σμίτση μπορεί να συνεχίσει να κάνει τα μπακλαβαδάκια της όπως αυτή το επιθυμεί. Το θέμα είναι λοιπόν να δούμε ε, τι θα γίνει με τις εταιρείες, οι μικροεπιχειρήσεις που ασχολούνται, εξαιρούνται σε περιόδους μέχρι πέντε έτη Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα να δοθούν περαιτέρω εξαιρέσεις γιατί διακρίνουμε το ένα πράγμα είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις και ένα άλλο πράγμα είναι τα, ε, οι μικρές. Τώρα για τα γεννητικά τροποποιημένα δεν ασχολούμεθα με το θέμα αυτό γιατί έχει γίνει αντικείμενο ρύθμιση σε κοινοτικό επίπεδο. Κάθε προϊόν το οποίο περιλαμβάνει γενετικά τροποποιημένα προϊόντα υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει ετικέτα Τώρα, για την μέθοδο σφαγής ζωικών προϊόντων για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους. Η πρόταση δεν ασχολείται με το θέμα αυτό. Έχουμε διακανονίσει την θρησκευτική σφαγή, τελετουργική σφαγή, με ένα κανονισμό που μόλις έγινε δεκτός και σχετικά με τις ετικέτες είναι μόνο στα πλαίσια εθελοντικών σχημάτων. Νομίζω ότι πάνω κάτω κάλυψα τις ε, παρεμβάσεις σας και περιμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια της συζήτησης. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον κύριο Ταραμπελά για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για όλα όσα είπατε. 13 νομίζω πήρα το λόγο. Ε, Κρέντιστη σίγουρα έδωσε αρκετές απαντήσεις όσον αφορά και τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. 1829 ο κανονισμός που αναφέρεται σε αυτά και για τη σφαγή είπατε εντελετουργική ότι είναι σε θελοντική βάση. Ωραία. Ε, για να δω. Εντάξει, δεν θέλω εδώ να ενοχλήσω κανένα, αλλά... Α, ναι, ας πάω στην κυρία Ρέμερς, σε μια παρατήρηση που έκανε εκείνη και η κυρία Ράμς, όσον αφορά τα αλκοπόψ αναφέρεται το αλκοόλ 7, 8 βαθμοί και 9 καμιά φορά. Ναι, αλλά αυτό που λέω είναι ότι επειδή τα πουλάνε με τα αναψυχτικά, σαν ένα αναψυχτικά, θα πρέπει να αναφερθεί και η ζάχαρη που είναι πάρα πολύ υψηλή η περιεκτικότητα σε ζάχαρη σε αυτά τα προϊόντα. Για μένα δεν ήταν τόσο το αλκοόλ που είχε πρόβλημα, όσο η περιεκτικότητα σε ζάχαρη, που σημαίνει ότι είναι προϊόν που δίνει πολλές θερμίδες. Τώρα ότι υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν δυσκολίες, αλλά είπα και πριν, υπάρχει βιομηχανία, υπάρχει διανομή, υπάρχουν οι παραγωγοί. Εγώ συναντήθηκα με καμιά εικοσαριά διαφορετικούς οργανισμούς και λόμπις και όταν έλεγα ότι θέλω να βάλουμε τον παραγωγό μου λέγανε «Μα ξέρετε, εμείς ε, τι, έχουμε μια αγορά παγκόσμια. Εμείς τις ντομάτες δεν ξέρουμε που θα αγοράσουμε τις ντομάτες μας. Σήμερα εδώ, μεθαύριο στην Κίνα ε, ναι, του λένε είναι παγκόσμια αγορά σα. Ε, εγώ θέλω καταναλωτή να ενημερώνεται για το πού αγοράζετε εσεί τι ντομάτε σα και για την ευρωπαϊκή αγορά. Δεν είναι για προστατευτισμό, αλλά είναι γιατί θέλουμε να παίρνουμε τα προϊόντα μα όσο γίνεται πιο κοντά σε εμά και για να ξέρουμε ποια είναι η ενέργεια που καταναλώνεται για να φτάσει το προϊόν μέχρι τον καταναλωτή. Ο καταναλωτή όλο και περισσότερο θα θέλει να το ξέρει αυτό. Και, χαίρομαι, και θέλω ε, οι πολυεθνικές μάλλον αγοράζουν από την Ιταλία την Ανταλουσία εξωγοπόλου στην Ευρώπη τις ντομάτες του παλού. Αν θέλουν να τις αγοράζουν στην Ταϊλάδη ή αλλού να τις αγοράσουν, αλλά να το ξέρουμε. Γι' αυτό προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Σίγουρα υπάρχουν περιορισμοί, αλλά αξίζει τον κόπο να το προσπαθήσουμε. Για τους σηματοδότες χαίρομαι που βλέπω. Κοιτάξτε, εγώ μίλησα για τους σηματοδότες εδώ, ενώ δεν το βάζω στην έκθεσή μου. Και γιατί, γιατί άλλες επιτροπές, η ΙΜΚΟ για παράδειγμα, το θέλουν. Η συγκήτρια είναι φίλη, αλλά το θέλει. Και εγώ ήθελα να σας το πω. Αν μπορούμε εμεί τις πολιτικές ομάδες να αντισταθούμε, τόσο το καλύτερο. Για το αλκοόλ λοιπόν είπα. Τι άλλο. Α, ναι, η πρωταρχική, το πρωταρχικό συστατικό παράρτημα 4, η πρώτη παράγραφος, και εδώ και η κυρία Γκοζίλα, εκτός αν γίνει Smith and Company. Αλλιώς δεν έχει σημασία το πρωταρχικό προϊόντο. Αν ε, μαγειρεύει τόσο καλά και τόσο πολύ, δεν μπορεί κάποια στιγμή να γίνει εν company. Εν πάση περιπτώσει, προς το παρόν πάντως το πρωταρχικό συστατικό πρέπει να είναι πάνω από 50%. Στο γλυκό που βάζει και λίγα καρύδια και λίγα πόλα είναι πιο δύσκολο. Ίσως να είναι το χαρακτηριστικό συστατικό. Μπορεί να είναι τα αμύγδαλα, μπορεί να είναι τα καρύδια. Αν είναι τρία, να βάζει και τα τρία. Ε, πιο πέρα δεν μπορούμε να πάμε, γιατί γίνεται υπερβολικά γραφειοκρατικό. Αλλά καταλάβαμε το βασικό συστατικό των προσυσκευασμένων υπάρχει. Αν είναι μπιζελόσουπα θα τα μπιζέλια. Και αν είναι ένα σύνθετο ε, τρόφιμο με σοκολάτα που είναι πάνω 5% είτε έρχεται από την ακτή ελεφαντος του Ιταλού, ξέρουμε ποιο είναι το πρωταρχικό συστατικό. Πάντως σας ευχαριστώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καλά δεν πρόκειται για την κυρία Σμιθ, αλλά το 3410 αναφέρεται στη μικρή κλίμακας παραγωγή και κάπου αλλού. Στο άρθρο όχι 16, ποιο είναι, τροπολογία 15, στο 45 που μιλάει για την ενίσχυση των μικρομεσαίων για τη μεταβατική περίοδο. Σίγουρα δεν πρέπει να τις ξεχάσουμε και να μην τις αναγκάζουμε να αντιμετωπίσουν τους ίδιους κανόνες που αντιμετωπίζουν και οι πολυεθνικές. Δεν θα μακρηγορήσω περισσότερο, θα συνεχιστεί η συζήτηση αναφίβολα. Περιμένω τις προτάσεις σας πάντως για τροπολογίες. Χαίρομαι πάντως που ήδη στο σύνολο της η έκθεση και όσον αφορά τις κύριες γραμμές πετυχαίνει συνένεση. Πραγματικά ιδιαίτερα που συζητήθηκε σήμερα που αρχίζει να ισχύει η Λισαβόνα. Καλώς και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με όλους τους συναδέλφους. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Μάρκ Ταλαμπερά για μια πολύ καλή δουλειά